So, dear colleague <laughs> and ladies and gentlemen, uh, let's start our... Oh, dear colleagues. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Έχετε ο καθένας ε, ημερήσια διάταξη, έχετε λάβει, έχετε λόγους να την αλλάξουμε, από ό,τι φαίνεται όχι, εγκρίνεται λοιπόν. Δεύτερο σημείο, έγκριση του σχεδίου πρακτικών ε, των συνεδριάσεων 20 και 21 Ιανουαρίου. Αν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης δεν υπάρξει αντίρρηση, θα θεωρηθεί ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Σημείο 3. Παρόμοια. Απόφαση, αποφάσεις των συντονιστών ε, του, του Ιανουαρίου, αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις ε, μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα, θεωρηθού, θα θεωρηθεί ότι έχουν εγκριθεί. Σημείο 4. Ε, η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται διαδικτυακά, είναι web stream. Καλώς ορίσετε λοιπόν όλοι οι ακροατές από το Ταλίν μέχρι τη Θεσσαλονίκη και φυσικά υπάρχει διερμηνία. Και Ζητώ από τους συναδέλφους να μιλούν σε λογικό ρυθμό και, με πάση περιπτώσει, όχι ταχύτατα. Σημείο 5. Η ενεξελίξη τριμερής διαπραγματεύσεις, μία διαπραγμάτευση στην ουσία, είναι η ο κανονισμός ε, ελέγχου εξαγωγών διπλής χρήσης ε, συνεδριάσεις της 13 Φεβρουαρίου. Η συνεδρίαση αυτή ήταν πολλά υποσχόμενη. Η Κροατική Προεδρία είναι πανέτοιμη να προχωρήσει και μοιάζει ότι υπάρχει και ένα περιθώριο ε, λιγμών από πλευράς Συμβουλίου. Έχει επέλθει πρόοδος στο θέμα της διαφάνειας, στο θέμα της υποβολής αναφορών, ε, αδειοδότησης και το σύστημα ε, αδειών γενικών εξαγωγών. Φυσικά, εξακολουθεί να υπάρχει θέμα στην αυτόνομη λίστα και το catch-all για τα θέματα της ε, πολιτικής τεχνολογίας και ακόμα και εκεί το Συμβούλιο έχει υποβάλει προτάσεις που αυτή τη στιγμή δεν μας αρκούν, αλλά και πάλι υπάρχει κάποια κίνηση. Παρίσταται και ο εισηγητής και θα του δώσω το λόγο για να κάνει συμπληρωματικά σχόλια. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ. Είπατε τα ουσιαστικά, Πρόεδρε. Είναι προτάσεις του Συμβουλίου. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη πρόταση. Μπορούμε να συζητήσουμε επ' αυτής της βάσης. Παλιά δεν συνέβαινε αυτό. Όπως είπατε και εσείς, χρειαζόμαστε και άλλες βελτιώσεις. Η Κομισιόν πρότεινε κάποια πράγματα τα οποία είναι αρκετά καλά αλλά όχι εντελώς. Είμαστε σε καλό δρόμο. Και ελπίζω ότι θα μπορούσαμε να τελειώσουμε το θέμα αυτό εν ευθέτω χρόνο. Ο επόμενος τριμερής διάλογος προβλέπεται να γίνει το Μάρτιο. Νομίζω στις 26 Μαρτίου, λέει ο Πρόεδρος. Στο μεταξύ έχουμε δύο τεχνικές συνεδριάσεις. Μπορεί να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία. Μπορεί. Στον επόμενο τριμερή διάλογο. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα. Μέχρι να συμφωνηθεί το πακέτο. Είναι ο χρυσό κανόνα των διαπραγματεύσεων. Ερωτήσει. Όχι. Πάμε στο 6. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Είναι η εφαρμογή της ε, εμπορικής πολιτικής μας. Πρόκειται για την ε, έκθεση για το θέμα αυτό. Και το μήνυμα, το σαφές αυτής της Επιτροπής, πέρα από την ε, συνάφεια, τη συνέπεια της πολιτικής, εστιάζουμε και, στις, και στην εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής, το πώς εφαρμόζεται και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ετοιμάσουμε τη δική μας έκθεση για την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής. Είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε μια τέτοια έκθεση εφαρμογής, η πρώτη φορά σε αυτή την νομοθετική θητεία και μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ένα πλατή προβληματισμό για τα θετικά και τα αρνητικά της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών το τελευταίο χρόνο. Και βεβαίως να δούμε τι θα γίνει και ποια στοιχεία χρειαζόμαστε να λάβουμε υπόψη μας για την ε, εφαρμογή της μελλοντική εμπορικής πολιτικής και των μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών. Ο κύριος Γουόρμπορν ε, θα, θα πάρει το λόγο για το πολύ πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι η ετήσια έκθεση πρωτοβουλίας για την εφαρμογή της κοινή εμπορικής πολιτικής. Είμαστε τώρα στη φάση σύνταξής της και η εξέτασή της θα γίνει στην εδριασή μας του Μαρτίου. Έχουμε μια πρώτη τώρα ανταλλαγή απόψεων και είναι μια καλή ευκαιρία για να ακούσω τις απόψεις σας. Η Κομισιόν τα τελευταία τρία χρόνια έχει ετοιμάσει μια ετήσια έκθεση για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών και μια ανάλυση για τα πορίσματά τους και είναι η βάση για τη δική μας έκθεση. Όμως η κοινή εμπορική πολιτική είναι πολύ ευρύτερη από την εφαρμογή των συμφωνιών ελευθερών εμπορίου. Το Κοινοβούλιο έγραψε την τελευταία τέτοιου τύπου έκθεση το 2018 και ήταν ε, επειδή πέρυσι ήταν εκλογική χρονιά, δεν ετοιμάσαμε τέτοιου τύπου έκθεση. Σημαντικό σημαντικό στοιχείο της έκθεσης του 2018, μάλλον σημαντικά, τα σημαντικά στοιχεία, παραμένουν. Και τα επαναλαμβάνω, αλλά κάποια στοιχεία πρέπει να αλλάξουν το κείμενο του 2018 και να λάβουμε υπόψη μας και τις εξελίξεις στο μεταξύ. Στην έκθεση πρέπει να εστιάσουμε στις προτεραιότητες σε θέματα σχέσεων με τις ΗΠΑ, Κίνα, Αφρική, τον ΠΟΕ, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη και τις συνεχείς, συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις, καθώς και το ψηφιακό εμπόριο και το εμπόριο στις υπηρεσίες. Θεωρώ ότι ένα ελεύθερο εμπόριο με βάση τους κανόνες είναι ο καλύτερος τρόπος, ούτω ώστε η Ένωση να γίνει πιο ανταγωνιστική σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί και σε ανταγωνιστικότητα και σε ανάπτυξη και περισσότερες συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και λιγότερα εμπορικά εμπόδια θα πρέπει να είναι ο στόχος μας. Ο ΠΟΕ πρέπει να μεταρρυθμιστεί εκ βάθρων. Ε, πρέπει να δούμε τι γίνεται με, τον, με την πολυμέρεια, με τη δυνατότητά μας να συνεργαστούμε π.χ. με τις ΗΠΑ για να επιλύσουμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Διάφορες πρωτοβουλίες έχουν γίνει για να επιληθεί η έλλειψη σώματος προσφυγών στον ΠΟΕ και θα γίνει δουλειά μέχρι την Υπουργική στο Καζακστάν. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η Υπουργική επίσης. Επίσης θα μπορούσαμε να φτάσουμε πιο κοντά σε συμφωνία σε κάποιες τομεακές διαπραγματεύσεις όπως για την αλληλεία και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Κίνα συνεχίζει να δημιουργεί πρόβλημα, γιατί παίζει με διαφορετικού κανόνες από του υπόλοιπου, ενώ είναι μια αγορά πολλών ευκαιριών λόγω μεγέθους και λόγω ανάπτυξης. Για το Καναδά ε, και τη Σιγκαπούρη γράφω και δίνω αυτά τα παραδείγματα ε, τα τελευταία χρόνια, που είναι με, τα, με χώρες με τις οποίες ε, ως ο θα μπουν συμφωνίες σε εφαρμογή. Η εφαρμογή σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία θα είναι πολύ σημαντική για να δούμε το ποσοστό χρησιμοποίησης των συμφωνιών μας. Υπάρχουν παρόλα αυτά και άλλες συμφωνίες που δεν έχουμε υπογράψει, που θα πρέπει να ε, υπογράψουν πράγματος χάρη μια σημαντική διαπραγμάτευση και συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ζηλανδία και Ταϊβάν επίσης. Και θα πρέπει να επικυρώσουμε την ε, συμφωνία με το Μερκοσούρ. Οι εμπορικές μας σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να γίνουν ως να τον πιο στενές και να επωφεληθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτό. Έχουμε την, ε, το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη από την άλλη. Η σημαντική Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και επιπτώσεις της στο εμπόριο, που θα είναι οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικά ισορροπημένες. Με το εμπόριο μπορούμε να διαδώσουμε την ευημερία και τις ευρωπαϊκές αξίες. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι το εμπόριο στις υπηρεσίες και το ψηφιακό εμπόριο για την ευρωπαϊκή οικονομία. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σημαντικό να τις σκεφτόμαστε όταν νομοθετούμε και να μην σκεφτόμαστε μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ζητώ από την Κομισιόν να τελειώσει τη δουλειά της για τους κανόνες προέλευσης και το εργαλείο αυτοαξιολόγησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να δει πώς θα εφαρμοστεί η αρχή one in one σε ό,τι αφορά την εμπορική πολιτική. Λόγω των περιορισμών, λόγω του μεγέθους της, μπορείτε να τη βρείτε πολύ σύντομη, αλλά καλύπτω μόνο τα σημαντικά θέματα. Και επειδή είναι η πρώτη φορά που στη νέα Επιτροπή ΙΝΤΑ ε, εκφράζουμε την άποψή μας για τα παγκόσμια εμπορικά θέματα. Θέλω να ακούσω τις απόψεις όλων των συναδέλφων. Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω το Ρέμι από τη Γραμματεία και τον Πιέρο από την ομάδα μας και την Κλάρα από τη δική μου ομάδα για την τεράστια βοήθεια που μου έδωσαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βόρμπαρν. Και τώρα να δώσω το λόγο στους και Ο κύριος Τάνας είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ και θα μιλήσω ισπανικά. Ευχαριστώ κύριε Warborn. Από το Renew θέλουμε να συνεργαστούμε. Περιμένουμε να βάλετε τα ακουστικά σας. Να προλάβει και η διερμηνία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Warborn. Ε, εξ ονόματος της Renew θέλουμε να συνεργαστούμε με όλου του συναδέλφου για να ετοιμάσουμε αυτήν την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2018. Ε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο εν το συνόλου τους. Πέρα από τα ε, ωφέλη του ε, διεθνούς εμπορίου, είναι πάρα πολύ ε, μέσω αυτών των συμφωνιών να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια και, τις, ε, και τους κανόνες. Ε, το θέμα είναι πώς εμπορευόμαστε σήμερα. Ξέρουμε ότι κάποια αξιώματα γύρω από το, εμπορι... από το διεθνές εμπόριο ε, αμφισβητούνται. Πολλοί πολίτες μας δεν θεωρούν, δεν αντιλαμβάνονται ότι το εμπόριο είναι θετικό, ότι δεν αυξάνει την ευημερία. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και μερικές φορές το εμπόριο τους ε, επηρεάζει αρνητικά. Αυτοί δεν επωφελούνται από τα ωφέλη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ ριζοσπαστικά. Τι θα πρέπει να ανανεώσουμε, ποιες αξίες, ποια αξιώματα, ποιες αρχές ε, θα πρέπει να αλλάξουμε για το εμπόριο, γιατί το εμπόριο ουσιαστικά είναι εκ των όνου κάνευ για, την, για το καλό και την ευημερία της ε, κοινωνίας μας. Και θα πρέπει βεβαίω να παρακολουθούμε την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής για να εντοπίζουμε και να εφαρμόζουμε μέτρα. Γνωρίζουμε ότι οι πολίτε έχουν ανησυχίες πολλαπλές για τις αρνητικές συνέπειες που έχει το εμπόριο στο περιβάλλον, ε, υπάρχει μία αποκοπή των πολιτών και οι εμπορικές συμφωνίες, παρότι μας βαραίνει αυτό, θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε και ανανεώσουμε τη συζήτηση για το εμπόριο και να λάβουμε υπόψη μας ανησυχίες των πολιτών. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε το αφήγημα γύρω από το εμπόριο και τη σημασία του. Και να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι εκ των όνου κάνευ για την ευημερία των χωρών μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, θα πρέπει να, σε αυτό που κάνουμε να εμπλέξουμε τους πολίτες, να τους φέρουμε κοντά. Και θα πρέπει να τους ενημερώσουμε για την εμπορική πολιτική ε, της Ένωσης και για το πώς εφαρμόζεται. Θα πρέπει να, να καταλάβουν οι, πολίτε οι πολίτες το εμπόριο, ε, ότι είναι πρόοδος, ότι είναι ανάπτυξη, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να είναι για όλους. Αυτή λοιπόν είναι η ανησυχία μας και γι' αυτό λοιπόν θέλω να δουλέψουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Muchas gracias. And the other shadows... Από τους και άλλες δεν βλέπω να είναι κανείς εδώ. Και δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο. So perhaps from my side... Από πλευράς μου λοιπόν τότε να κάνω κάποια σχόλια. Είπατε και δίκιο είχατε ότι ο βαθμός χρήσης στις εμπορικές συμφωνίες είναι αρκετά χαμηλός. Και αυτό θα πρέπει να το βελτιώσουμε, να δούμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθεί πιο πολύ αυτές οι συμφωνίες από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα μεγάλο βήμα και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα προωθήσουμε αυτές τις νέες δυνατότητες. Για να υπάρχει πραγματικά όφελος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και κατά δεύτερον, αν σωστά καταλαβαίνω από την έκθεση, έχουμε και κάποια μεμονωμένα μικρά στοιχεία επί των οποίων διαφωνούμε με τους εταίρους μας. σε ό,τι αφορά τους κρατικούς φορείς για την Κορέα, για παράδειγμα την επικύρωση του σκέλους για τα εξαρτήματα αυτοκινήτων στην Νότια Κορέα. Άλλα στοιχεία σε ό,τι αφορά την Ιαπωνία. Και αναρωτιέμαι για το κατά πόσον μπορεί να υπάρξει κάποια σαφής διαδικασία για να βελτιωθούν οι λεπτομέρειες των συμφωνιών αυτών. Προκειμένου τα προβλήματα αυτά να μην συνεχίσουν να εμφανίζονται και σε εμπορικές συμφωνίες. Για παράδειγμα, τέθηκε ένα θέμα για τη χρήση των ποσοστώσεων ιδιωτήρη στον Καναδά. Υπάρχουν λοιπόν σε κάποιες περιπτώσει κάποια παρατηράκια τα οποία πραγματικά θα πρέπει να βρούμε τρόπο να τα κλείσουμε. Αυτά ήταν τα σχόλιά μου. Και άλλα δύο σχόλια έχουν να κάνουν, έχουν να κάνουν συναδελφοί καταρχά από την κυρία Ροντρίκη Σπινιέρο. Ευχαριστώ. Για το σημείο 6. Και για τα όσα είπε ο εισηγητής για αυτό το, το θέμα, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση και να πω μία σειρά επιχειρημάτων. Καταρχάς για την ερώτηση. Το εμπόριο με τις τρίτες χώρες, όταν έχουμε συμφωνήσει ελευθέρου εμπορίου, ε, αναπτύσσεται λιγότερο από το εμπόριο με τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν έχω δει ανάλυση όμως γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι γιατί οι χώρες αυτές ζητούν λιγότερο τα προϊόντα μας, υπάρχει δυσκολία πρόσβασης, δεν καταλαβαίνω. Θα ήθελα να δω κάποια αναλυτικά στοιχεία για την ε, εξέλιξη που έχει παρουσιαστεί αυτή και που μας παρουσίασαν. Επίσης, για το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό το κεφάλαιο δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένο στην έκθεση που μας παρουσίασαν. Θα ήθελα περισσότερα στοιχεία. Πάντως θεωρούμε ότι είναι θετικό το, το γεγονός ότι γίνεται αυτή η αξιολόγηση και αυτή η ανάλυση που δεν μπορούσε να γίνει το 2019 λόγω εκλογών. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να γίνεται, όπως είπε και ο συγητής για να το αναλύσουμε πώς θα βελτιώσουμε την ε, εφαρμογή των συμφωνιών και την ε, διαπραγμάτευση νέων συμφωνιών. Η ομάδα μου ενδιαφέρεται πάρα πολύ για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του κεφαλαίου της βιώσιμης ανάπτυξης και να περιλαμβάνει πάντα την κοινωνική ευθύνη και την εταιρική ευθύνη, να βάλει ειδικά κεφάλαια για το φύλλο το 21ο αιώνα δεν μπορούμε να υπογράφουμε εμπορικέ συμφωνίε που δεν λαμβάνουν υπόψη την προοπτική του φύλου και την ειδική θέση που βρίσκεται ο μισός πληθυσμό. Επίσης μας φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό η συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, να λαμβάνει υπόψη από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ποια είναι η θέση που θα προτάξουμε, θα προτάξει η Κομισιόν για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να μάθω παρακαλώ. Ευχαριστώ. Uh, και τώρα. Μπορέλ. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη από τον εισηγητή. Ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Και προφανώς ε, ε, αυτό που θέλουμε να επιτύξουμε είναι ότι η εμπορική πολιτική τη της Ευρωπαϊκής είναι καλή και είναι καλή και η ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων και αγαθών. Μία παρατηρήση να κάνω όμως. Σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες, ε, ε, τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, επ' αυτού συμφωνούμε, αλλά είναι δύο τομεί όπου διαρκώ παρουσιάζεται πρόβλημα ανάπτυξη βιώσιμη ή τα κοινωνικά ζητήματα. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, στην Νότιο Κορέα. Εξαιρετικά τα θέματα σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας αυτής, αλλά Όντω, η Νότια Κορέα δεν έχει επικυρώσει μία σειρά συμβάσεων και πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βρίσκεται στην ε, θέση να ζητάει από την Νότια Κορέα να επιταχύνει και την ίδια συζήτηση έχουμε και το Βιετνάμ σε ό,τι αφορά τα ανθρωπίνα δικαιώματα και σε 3-4-5 χρόνια οι διαδοχή μα θα έχουν ακόμα τι ίδιε συζητήσει ε, με την Νότια Κορέα. Σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, βρισκόμαστε σε μια φάση όπου διαπιστώνουμε ότι α, καλά πάνε τα πράγματα γενικά, αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά τα φυτοπροστατευτικά, το περιβάλλον κτλ. Αυτό ισχύει και με την ΣΕΤΑ και στις 17 Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από μία ΜΚΙΟ σε ό,τι αφορά τι ε, επιτρόπους, σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία και στην έρευνα αυτή αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά του Καναδά και στα ευρωπαϊκά φόρουμ κτλ. ότι υπάρχει απόπειρα να αμφισβητήσουν τα φυτοπροστατευτικά μας μέτρα. Άρα εμείς ε, είμαστε περήφανοι για τις εμπορικές αυτές συμφωνίες, αλλά για τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά ζητήματα δεν είμαστε σε καλό επίπεδο. Θα, θέλαμε λοιπόν να ζητήσουμε την Επιτροπή να αλλάξει αυτή η στάση. Ευχαριστώ, κύριος Χάνσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω και το Γιούργεν για το τεράστιο έργο, την τεράστια δουλειά που έχει κάνει ως τώρα και για την πολύ εκτενή παρουσίαση, γιατί πολλά στοιχεία τα ακούσαμε ήδη. Δύο μόνο θέματα θα ήθελα να προσθέσω σε ό,τι αφορά το PIT με την Ταϊβάν. Εδώ η δική μας επιτροπή έχει πολύ έντονη τοποθέτηση. Το έχουμε αναφέρει σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν. Ίσως θα μπορούσαμε να το προσθέσουμε, ίσως και να το έχετε βάλει κάπου και να μην το έχω δει, γιατί δεν διάβασα ακόμα την έκθεση δυστυχώς αλλά είμαι σίγουρο ότι αυτό θα μπορούσαμε να το περιγράφουμε. Και θα θέλαμε να είμαστε πιο ακριβείς και λεπτομερείς ό,τι αφορά τους ε, κανόνες περί Γιατί η Επιτροπός ε, Μάλμστρεμ τότε απάντησε ταχύτατα στην ερώτησή μας. Ε, μετά από μια εβδομάδα απάντησε στην γραπτή μας ερώτηση και Αναφέρεται ότι πλέον δεν αναφέρεται ως rules of origin, αλλά access to market platforms, πρόσβαση σε πλατφόρμες αγορών. Και ότι θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία αρχές του 2020. Με φτάσαμε αρχές 2020. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε και να ασκήσουμε πιο πολλές πιέσεις και να δούμε τι ημερομηνίε μας έχουν υποσχεθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ρέγκη Μίντι από το ID έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα που συζητάμε για την ενεργοποίηση της κοινή εμπορικής πολιτικής μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε απολογισμό για τις πιο σημαντικές εμπορικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε. Όπως ε, τόνισα και χθε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Υγείας κατά την ανταλλαγή απόψεων με την ε, αρμόδια Επίτροπο, θα ήθελα να εκφράσω τα προβλήματα που έχω για την συνέπεια της ε, ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής με τους φιλόδοξους, σε σχέση με τους φιλόδοξους στόχους που έχει η σημερινή Επιτροπή για το περιβάλλον, την υγεία, την διατροφική ασφάλεια των πολιτών μας. Ιδίω, νομίζω ότι δεν μπορούμε ενσυνείδητα να μιλάμε για διατήρηση της ε, βιοπικιλότητας όταν χρησιμοποιούμε ε, φυτοφάρμακα και να δεχόμαστε ότι εισάγουμε τεράστιες ποσότητες από τρίτε χώρες, οι οποίες δεν είναι ευθυγραμμισμένε με τα ευρωπαϊκά μας πρότυπα. Επίση, δεν μπορεί η Ευρώπη σε καμία περίπτωση να καταπολεμήσει αποτελεσματικά τον καρκίνο και παράλληλα να ανοίγει ε, το εμπόριό της σε καρκινογόνες ε, ουσίες ε, και σε ενδοκρινικούς διαταράκτες που έρχονται μαζί με προϊόντα τρίτων χωρών. Θέλω ως Κοινοβούλιο να πάρουμε μια δυνατή θέση, ούτως ώστε να βάλουμε ένα φρένο στην, στον αθέμητο ανταγωνισμό ε, που μπαίνουν ε, προϊόντων που μπαίνουν στην αγορά μας χωρίς να σέβεται, σέβονται τίποτα, χωρίς να σέβεται τον ανταγωνισμό και θα πρέπει οι δικές μας πολιτικές να εφηγρομίζονται με τις επιτροπές αυτές, με τις πολιτικές των τρίτων χωρών. Ε, περιμένουμε το σχέδιο έκθεσης για να δουλέψουμε επικοδομητικά και να φτάσουμε σε μια λογική κοινή θέση. Ευχαριστώ. Thanks. Um, and now from the Commission Την κυρία Γεραλντίν Μέργκερ έχουμε τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να μας πει δύο λόγια και σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των κανόνων προέλευσης και το πώς πάνε τα πράγματα. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την εκ νέου πρόσκληση. Είναι πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση καθώς έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία της τέταρτης έκθεσης που θα δημοσιευτεί στο τέλος της χρονιάς. Είναι πολύ επίκαιρη η συζήτηση και όλες οι παρατηρήσεις σας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. Φυσικά είμαστε σε μια σημαντική συγκυρία όπως είπατε. Η προηγούμενη Επιτροπή σύναψε περίπου 15 νέες συμφωνίες που αντιστοιχούν αυτή τη στιγμή στο 31% του εξωτερικού εμπορίου της Ένωσης όταν θα ολοκληρωθούν όλες οι διαπραγματεύσεις θα αντιστοιχούν στο 50, 45% του εξωτερικού εμπορίου. Άρα είναι πολύ σημαντικό η παρούσα Επιτροπή να ασχοληθεί με την ε, εφαρμογή του FTA. Και βεβαίω ο υπεύθυνο για αυτά θα είναι στο επίκεντρο της προσπάθειας. Τώρα, αν δούμε την έκθεση, Είπε κάποιος συνάδελφος ότι ο σκοπός είναι να προωθηθούν οι FTA και η πολιτική της Κομισιόν για το εμπόριο. Όμως νομίζω ότι για μένα είναι μια ευκαιρία να επισημάνουμε τι λειτουργήσε καλά και τι δεν λειτουργήσε καλά και να επιδιώξουμε να βελτιώσει η κατάσταση. Αναφερθήκατε στο γεγονός ότι η συμφωνίες ε, συνεισέφεραν στην βελτίωση των, ε, του εμπορίου εισαγών και εξαγωγών, αλλά οι φυστάμενες όπως η ΣΥΤΑ και αυτή με, τις, ε, με την Ιαπωνία που τα πράγματα πάνε καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, όπως επίσης και το γεγονός ότι οι εμπορικές συμφωνίες μας βοήθησαν να αντιμετωπίσουμε τα εμπορικά εμπόδια και να προλάβουμε την δημιουργία τους. Επίσης υπάρχουν και κάποια παραθυράκια τα οποία εντοπίστηκαν και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ένα είναι φυσικά η χρήση των εμπορικών συμφωνιών και όταν πρόκειται για αγορά αγαθών είναι η χρήση των προτιμήσεων το ποσοστό χρήσης προτιμήσεων είναι ένας αδρός δείκτης και παραμένει τέτοιος γιατί η Κομισιόν τα ποσοστά τα υπολογίζει επί τη βάση των στοιχείων των στατιστικών των ε, τελωνιακών αρχών της κάθε χώρας. Είναι διαφορετικές οι μέθοδοι και άρα είναι πολύ ε, δύσκολο λοιπόν να συγκριθούν οι, τα ποσοστά χρήσης της Αιγύπτου και της Κορέας. Και ε, Βεβαίω ε, είναι διαφορετικό, είναι δύσκολο να συγκριθούν οι χρονιές το 17, το 18 και το 19 γιατί τα πακέτα είναι διαφορετικά. Τι κάνουμε λοιπόν, ε, κινούμαστε σε διάφορα μέτωπα. Πρώτον, προσπαθούμε όλο και περισσότερες χώρες να στείλουν δεδομένα. Το 2019 πήραμε ε, 26 σειρές δεδομένων. Έχουμε νέα συμφωνία που να περιλαμβάνουν διατάξεις που υποχρεώνουν τους εταίρους να υποβάλουν στοιχεία περιοδικά. Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις για να δούμε γιατί κάποιοι δεν χρησιμοποιούν τις προτιμήσεις ακόμα και επίσης, πολύ σημαντικό, ε, προετοιμάζουμε ε, μια νέα πύλη, ε, μια νέα διαδικτυακή πύλη που θα διευκολύνει τη χρήση και την πρόσβαση σε φιλική προς το χρήστη πληροφορία. Και επίσης κατά τον Απρίλιο ή Μάιο μαζί με την νέα Chief 24 θα υπάρχει ένας ε, ένα ε, εργαλείο αυτό των κανόνων προέλευσης ε, θα, χρησιμοποιηθούν, θα χρησιμοποιηθεί από πολλές εταιρείες. Εμεί τι προσπαθούμε. Προσπαθούμε να πετύχουμε ένα δένδρο λήψη αποφάσεων και να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένες αποφάσεις, ξεκινώντα από τι πιο πρόσφατε, όπως αυτή με την Ιαπωνία και τη ΣΥΤΑ, και να προχωρήσουμε για να υπάρχει μια διαδραστικότητα και να μπορέσουν να καλυφθούν διάφορα πεδία. Οπότε να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες ε, για το εάν και κατά πόσον ένα προϊόν πιθανώς θα, ε, θα συμμορφώνεται με τους κανόνες προέλευσης και θα υπάρχει ωφέλεια από αυτό. Επίσης όλα αυτά θα τα δοκιμάσουμε με τους χρήστες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις και θα υπάρχει διαρκής βελτίωση. Όταν θα ξεκινήσει αυτό θα ε, διαπιστωθεί ότι θα υπάρξουν πολλές βελτιώσεις στην πρόσβαση ε, στις πληροφορίες, αρκετά καλού επίπεδου μηχανική μετάφραση σε διάφορες γλώσσες και ένα εργαλείο ε, και πολλές περισσότερες πληροφορίες για διάφορες FTA. Ε, Έτσι θα υπάρχουν επίσης δραστηριότητες προώθησης σε κράτη-μέλη. Όλα αυτά είναι στη φάση προετοιμασίας. Αναφέρθηκαν και τα ποσοστά του τυριού, ποσοστός τυριού για τον Καναδά, ε, το πρόβλημα με τα πρότυπα των αυτοκινήτων στην Νότια Κορέα. Αυτά τα ε, παραθυράκια εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα και μετά τη σύναψη FTA. Ε, καταρχήν, όταν έχουμε μια πρόσφατη τέτοια συμφωνία, διαπιστώνουμε ότι η ερμηνεία κάποιων άρθρων αυτής της συμφωνίας διαφέρουν από τη δική μας πλευρά και από την πλευρά της, των χωρών εταίρων. Τι κάνουμε λοιπόν στις επιτροπές και σε τεχνικό επίπεδο αλλά και στην ανώτατο επίπεδο θέτουμε θέματα όπως τα ποσοστά του τυριών, των τυριών. Ας πούμε Είχαμε την περίπτωση της Ιαπωνίας. Είπαμε το θέμα της ερ, ερμηνείας των κανόνων προέλευσης και ότι πρέπει οι επιχειρήσεις να μπορούν να επωφελούνται από αυτούς τους κανόνες. Αυτό το κάνουμε στις επιτροπές. Προσπαθούμε να ε, έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια στο, ε, για το αποτέλεσμα αυτών των ε, ε, επαφών και ε, αναβάζουμε στην ιστοσελίδα μας την ημερήσια διάταξη και τις αναφορές για τις επιτροπές. Κατά τα λοιπά είμαστε σε διαρκή ε, διάλογο με τη, τους εταίρους μας για να τους πείσουμε να αναρτήσουν τα προϊόντα αυτά στην ιστοσελίδα. Τώρα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, όντως είναι ένα σημαντικό θέμα τα θέματα αυτά έχουν εξελιχθεί, τα TST, από τότε που ξεκινήσαμε με την Νότια Κορέα για πρώτη φορά, τα εξετάζουμε όλα αυτά στο πλαίσιο της εκτονιστέρων των υστέρων αξιολόγησης. δημοσιεύτηκε η εκ αξιολόγηση με την Κορέα, μετά ε, με τις χώρες Κεντρικής Αμερικής, τις χώρες της κοινότητας και για τις χώρες της Μεσογείου θα υπάρξει ένας πρώτος διάλογος κοινωνίας των πολιτών τον Μάρτιο Προσπαθούμε λοιπόν και να βρούμε άλλους τρόπους να ε, συνεργαστούμε ε, για θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπήρξαν και άλλα ζητήματα που ετέθησαν, όπως συγκεκριμένα γιατί ε, πέρσι, όχι το πρόπερσι, αλλά πέρσι αναπτύσσεται πιο αργά το εμπόριο στο πλαίσιο των FTA πρέπει να πω το εξής. Πρώτον, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο και περιβάλλον και τις εντάσεις, ε, τους εμπορικούς περιορισμούς, καθώς και άλλα στοιχεία. Αναφέρθηκα μεγάλη συντομία όταν παρουσίασε την έκθεση ότι υπάρχουν στην Τουρκία, ας πούμε, εμπορικοί περιορισμοί όπου έχουμε δει ε, αύξηση των εμπορικών ε, εμποδίων και επίσης το εμπόριο με τη Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιστοιχεί στο 30 περίπου Οπότε ε, όταν αυξάνεται από εκεί, το πράγμα που μας αρέσει, έχουμε μείωση αλλού. Θα έχουμε περισσότερη ανάλυση στην επόμενη έκθεση. Ε, ήδη, ζητώ συγγνώμη. Στο σημείο αυτό θα κλείσω και προσβλέπω στην συνέχιση της συνεργασίας μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Θα προσπαθήσω όσο καλύτερα μπορώ να ε, δουλέψω. Υπάρχουν πολιτικές δυσκολίες και σε μερικές περιπτώσεις τα πράγματα είναι πιο εύκολα, σε άλλες πιο δύσκολα. Υπάρχει ένα θέμα που εκρεμεί από αυτά που είπε ο κ. Κάνιες, ο οποίος με μεγάλο πάθος αναφέρθηκε στην αντίληψη από πλευράς των πολιτών ε, στην αντίληψη του εμπορίου από τη σκοπιά των πολιτών. Πρέπει να πούμε ότι όλο και περισσότερο ο κόσμος διαπιστώνει τα ωφέλη του εμπορίου, ε, πολύ περισσότερο από ότι την προηγούμενη φορά που έγινε μια έρευνα. 60% τώρα ε, ε, ε, αισθάνονται ότι ωφελούνται προσωπικά από το διεθνές εμπόριο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει ανέβει το ποσοστό κατά 16 μονάδες. Μερικές φορές διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά όσο είναι στην πραγματικότητα. αντιλαμβανόμαστε μάλλον τα πράγματα λιγότερο καλά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και αυτό θα το αναφέρω, το, το στοιχείο θα το αναφέρω στην έκθεση και θα συνεργαστώ με τον κύριο Κάνιας για να βρούμε τρόπους ε, ώστε να γίνει ε, προσπάθεια να αυξηθεί τώρα το, το, ποσοστό αυτό. Ε, χρονοδιάγραμμα. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα εξεταστεί το Μάρτιο το πρώτο σχέδιο έκθεσης. Η προκαταρτική μου έκθεση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη ε, θα σας ζητήσω να τη διαβάσετε και να σχολιάσετε και βεβαίως θα υπάρξουν ε, προθεσμίες για υποβολή τροπολογιών μετά την επόμενη συνεδρία του Μαρτίου, 24 Μαρτίου. Ευχαριστώ και πάλι πολύ για τα σχόλιά σας. Λοιπόν, ε, Ευχαριστούμε κύριε Βόρμπον. Τελειώνουμε έτσι με το σημείο 6 και θα περάσουμε στο 7. Είναι μια ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας για παραχωρήσεις για το κρέας. Ο, ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Warborn. Ξανά. Του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση είναι η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου να συμφωνήσει το Συμβούλιο για παραχωρήσει της Ελβετίας στον ΠΟΕ για τον κρέας που δεν έχει υποστεί άλλη επεξεργασία πέραν του καρικεύματος. Οι δεσμολογικές ποσοστώσεις για το καρικευμένο κρέας ε, ήταν είναι χαμηλότερες από το μη καρικευμένο κρέας και ορισμένοι εισαγωγοί το παρέκαψαν αυτό βάζοντας αλάτι στο κρέας ας πούμε και πιπέρι ε, πριν από τα σύνορα και μετά ξεπλένοντάς το αφού μπει το κρέας στην Ελβετία. Το 2015 το Κοινοβούλιο της Ελβετίας ε, αποφάσισε να αυξήσει αυτές τις δεσμολογικές ποσοστώσεις για να, για να αντιμετωπίσει έτσι τις αυξανόμενες εισαγωγές. Αυτό μπήκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2016. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος και προσπάθησε να το λύσει διμερώς. Και τελικά το 2017 η Ένωση αναγκάστηκε να προσφύγει στον ΠΟΕ για δράση, προσφεύγοντας τον ΠΟΕ και λέγοντας ότι δεν είναι συμβατό με τους κανόνες του ΠΟΕ. Η Ελβετία ξεκίνησε μια διαδικασία για να αλλάξει την παραχώρηση της ε, στον, προς τον ΠΟΕ. Επιτρέπεται αυτό από τον ΠΟΕ μετά από διαπραγματεύσεις και συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα μέλη μέρη, ας πούμε, και, κυρίως, και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη εδώ. Η λύση ήταν συμφωνία μέσω ανταλλαγή επιστολών να αυξήσουν τις ε, τεχνολογικές ποσοστώσεις, τους δασμούς για το καρικευμένο κρέας από από 791 ε, ευρώ ε, ανά 100 κιλά στα 2.043 ευρώ. και η δασμολογική ποσόστοση αυξάνεται κατά 12.000 τόνους. Επομένως, η Ένωση παίρνει ένα δασμό που αποκαθιστά την, την προηγούμενη πρόσβαση για το καρικευμένο κρέας στην αγορά της Ελβετίας. Η διμερή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας δεν έχει αλλάξει, αλλά με βάση με την κοινή εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η συμφωνία παρόλα αυτά απαιτεί την σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ένα πολυτεχνικό θέμα και συστήνω στο, στην ομάδα μας, στην Επιτροπή μας, να δώσει τη σύμφωνη γνώμη της. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανένα από τους σκιώδες να είναι εδώ. Η καρινα έχει να κάνει κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ. Δυστυχώς η συνάδελφός μου δεν μπορεί να παρευρεθεί στην συνεδρίαση σήμερα. Θα μιλήσω λοιπόν εξ ονόματος του, ως τον αδελφός μου. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο καταρχάς για την έκθεση. Και από ό,τι ακούσαμε, η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελβετία είναι στενή και είναι σημαντική. Και είναι ιδιαίτερο σημαντική σε ό,τι αφορά το κρέας είναι βασικός ε, εξαγωγέας κρέατος προς την Ελβετία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό που υπάρχει αυτή η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση και Ελβετίας για να αποφευχθούν παραθυράκια και ο σκιώδη του Renew Europe υποστηρίζει να δοθεί έγκριση για τις προτινόμενες αλλαγές σε ό,τι αφορά την εντολή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Ζητά κανείς το λόγο. Όχι. Μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από, προς τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διευθυνσής Άγκρη. Εξ γνωρίζω, αυτό ήταν ένας προσωρινός ε, μια προσωρινή πρόταση χωρί την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό είναι πολύ ασυνήθιστο, γιατί είναι σαφεί ε, οι συμφωνίε μα με την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Δεν θα υπάρχει σε καμία περίπτωση προσωρινή εφαρμογή ε, συμφωνία χωρί την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ρωτώ λοιπόν, γιατί δεν ε, κάνει και η Γενική Διεύθυνση Άγκρη αυτά που κάνει η Γενική Διεύθυνση Trade. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και καλημέρα σα. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποια παρανόηση σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε. Δεν εφαρμόζονται προσωρινά η συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας δώσω και το συγκείμενο, το γενικότερο πλαίσιο. Πρόκειται μια επιτυχή αμα, ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τις ε, συναλλαγές με την Ελβετία, η οποία Ελβετία ο, αύξησε τις τιμές και πέρα από τις ε, υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στα πλαίσια του ΠΟΕ. Μετά από τη διαδικασία που κίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, ξεκίνησε και αποδέχτηκε επιτέλους η Ελβετία να, να διορθώσει τις τιμές αυτές. Μιλάμε για 20 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον δασμούς ανά στις εξαγωγές μας για να εξαγάγουμε τα προϊόντα μας προς την Ελβετία. Κάναμε λοιπόν διαπραγματεύσεις με την Ελβετία για τις ποσοστώσεις 1.200 τόνοι, 600 τόνοι για καρικευμένο κρέας και οι Ελβετοί αποδέχτηκαν να εισαγάγουν και με χαμηλότερη ποσόστοση κρέας το οποίο προορίζεται για μεταπίεση. Αυτό είναι ικανοποιητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να σας απαντήσω, αυτή η συμφωνία δεν περιλαμβάνει καμία υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υποχωρήσεις που γίνονται αυτηρά και μόνο από την ε, Ελβετία για να μας αποζημιώσουν για την αύξηση που έγινε στους δασμούς που ήταν ε, πάνω από το επίπεδο που είχαν συμφωνήσει στο, για τον ΠΟΕ. Δεν υπάρχει λοιπόν κάνει καμία υποχώρηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε πρόκειται να κάνει. Αυτό που προβλέπει μόνο η συμφωνία είναι ότι επιτρέπουμε στην Ελβετία να κλείσει στη Γενέβη, στον ΠΟΕ, την υπόθεση αυτή. Όταν θα γίνουν οι αλλαγές οι οποίες έχουν υποσχεθεί, που μα έχουν υποσχεθεί. Η Ελβετία, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία, θα έπρεπε να ζητήσει επικύρωση τη συμφωνία ε, στη Γενέβη πρωτού εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά. Αυτό μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο. Αλλά μονομερός έχει αποφασιστεί από 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτου να ε, εφαρμοστούν αυτέ οι αποζημιώσει Ακόμα και αν αυτέ οι διαδικασίε σε επίπεδο που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα εγκαίρω. Δεν υπάρχει λοιπόν οποιοδήποτε θέμα σε ό,τι αφορά την προσωρινή εφαρμογή τη συμφωνία αυτή και ιδίω όχι από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που έγινε ήταν το εξή. Μονομερό η Ελβετία, και αυτό πρέπει να μα ικανοποιεί, αποφάσισε να μα δώσει την αποζημίωση αυτή, ακόμα και ενδεχομένω πιο πριν από την στιγμή που θα είναι νομικά υποχρεωμένη να το κάνει αυτό. Αυτό είναι προφανώ προ το συμφέρον των εξαγωγέων μα, οι οποίοι σήμερα ακόμα πληρώνουν 20 εκατομμύρια επιπλέον δασμού ανά έτο. Είναι θετικό, λοιπόν αυτό και τονίζω, το υπογραμμίζω εκ νέου. Δεν υπάρχει καμία, κανένα θέμα ότι αυτή η συμφωνία θα εφαρμοστεί προσωρινά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο μέχρι ότου συνενέσει το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις. Είναι λοιπόν το θέμα από πλευράς Ελβετίας ε, μια μονόπλευρη, ένα μονόπλευρο βήμα. Ευχαριστούμε πολύ ε, για την δέσμευση της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη, χωρίς, η οποία δεν θα δώσει καμία έγκριση χωρίς τη συνένεση του ε, Κοινοβουλίου. Κύριε Βόμποκ, δεν έχω τίποτα να προσθέσω στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Οπότε, 25 Φεβρουαρίου είναι η τελική ημερομηνία υποβολής προ, ε, τροπολογιών, ψηφοφορία στις 17 Μαρτίου. Ευχαριστούμε. Σημείο 8 τώρα. Γνωμοδότηση της ΑΦΕΤ για την Ανατολική Εταιρική Σχέση εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου εισηγητής η κυρία Μαρκέτα Γρεγορόβα των Πρασίνων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχω έρθει να παρουσιάσω το σχέδιο ε, γνωμοδότησης, σύστασης για την ε, Επιτροπή, το Συμβούλιο, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου, σε σχέση με την ετονική εταιρική σχέση. Στην εταιρική σχέση εμπλέκονται έξι χώρες, η Αρμενία, ε, Αζερβαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδοβία, Ουκρανία και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2019 γιορτάστηκε η δέκατη επέτειο Τη της ανατολικής εταιρικής σχέσης και απεδείχθη ότι η συνεργασία είναι ε, αμοιβαίως επωφελής, είναι κομμάτι μιας πολιτικής που σκοπό έχει την στενή, στενότερη σύνδεση, την οικονομική ολοκλήρωση και τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για ε, ε αντιμετώπιση κοινών ε, προκλήσεων όπως ας πούμε η βιώσιμη ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή. Υπάρχει διμερή συνεργασία και χρειάζεται να τονίσουμε τη σημασία της αμοιβαία συνεργασία. Εδώ υπογραμμίζω την σημασία της πλήρους υλοποίησης των συμφωνιών και ζητώ από την Ένωση να ε, ε, εξασφαλίσει ότι δεν θα παραβιάζονται οι στόχοι της κλιματικής αλλαγής και, τους, ε, ε, της, και του Green Deal. Οι, οι προϋποθέσεις της μικροοικονομικής βοήθειας είναι πολύ σημαντικές. Η βοήθεια που ε, προσφέρει η Ένωση πρέπει πάντοτε να συσχετίζεται με δημοκρατισμό και μεταρρυθμίσεις για να εξασφαλιστεί η σταθεροποίηση της γειτονίας που θα παραμείνει στις αρχές και τις αξίες της. Εξακολουθώ να ανησυχώ για θέματα διαφθοράς διαφθοράς και διακυβέρνησης μεταξύ των οποίων και η φοροδιαφυγή. Πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ζητώ την συνέχιση της, ε, της ε, χρηματοδότησης, ζητώ από την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της χρηματοδότησης και υπογραμμίζω την ανάγκη να μην απομακρυνθούμε από τις προϋποθέσεις για τον εκδημοκρατισμό και τις μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, βοηθώ για τη βοήθεια, ε, την βελτίωση του σχεδίου και βεβαίω προσβλέπω στη συνεργασία των σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ. Το λόγο έχουν οι σκιώδης εισηγητέ από το ε, ΕΛΚ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι θα προσπαθήσω ε, να μην επαναλάβω αυτά τα οποία είπε η εισηγήτρια γιατί η γνωμοδότησή της είναι πολύ ολοκληρωμένη, σύντομη αλλά πολύ έντονη ε, όσον αφορά την ουσία. Ε, η ανατολική εταιρική σχέση που ξεκίνησε το 2009 ε, ξεκίνησε ως πρωτοβουλία ειρήνης και δεν ε, έχει στόχο κανέναν. Αυτό είναι κάτι που θέλω να το υπογραμμίσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει ε, συμφωνίες σύνδεση με ε, την Μολδαβία, τη Γεωργία και την Ουκρανία και εκατόπιν ε, συμφωνίε με την Αρμενία, τη Γεωργία και το Αζερβατζάν και έχει ξεκινήσει μια διαδικασία με τη Λευκορωσία. Η εταιρική μας σχέση έχει εξελιχθεί ε, στη διάρκεια, στο πλαίσιο δύσκολων γεωπολιτικών συνθήκων και ε, έχουν υλοποιηθεί πολλές συμφωνίες. Εμείς εδώ ως ΙΝΤΑ πάντοτε επικεντρωνόμασταν στους ανθρώπους και την στενή συνεργασία μεταξύ πολιτών και ψηφίζαμε υπέρ των ε, ε, εταιρικών σχέσεων και των εμπορικών σχέσεων που τους τις υποστηρίζουν. Άρα είναι ευπρόσδεκτο αυτό το πλαίσιο το οποίο δημιουργήθηκε την διάσκεψη κορυφής ε, της ε, Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στην Ρήγα είναι το 2014 είναι ε, ευπρόσεπτες οι είναι πρόσδεκτοι στόχοι. Η ενίσχυση της ε, ε, ε, καλής διακυβέρνησης, η συνδεσιμότητα, η κλιματική αλλαγή, η κινητικότητα, οι επαφές μεταξύ των λαών και πολλά άλλα. Το ΕΛΚ στηρίζει την ε, ε, ε γνωμοδότηση που παρουσίασε η συγγήτρια κυρία Γκρεγορόβα για την οικονομική ολοκλήρωση των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Υπογραμμίζουμε τη σημασία της πλήρους υλοποίησης των ε, εμπορικών ε, ε, των συμφωνιών εμπορικού, ελευθέρου εμπορίου μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Σχέσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για επιχειρήσεις και εμπορικές ανταλλαγές. Όμως πρέπει να υποστηρίξουμε την για τις χώρες της Ανατολικής εταιρικής σχέσης να ε, έχουν περισσότερη βοήθεια από πλευράς Ένωσης για την διακυβέρνηση και την στήριξη οικονομικών μεταρρυθμίσεων και των ε, χρηματοοικονομικών τομέων και του δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρει μικροοικονομική ε, βοήθεια της Ένωσης για την ανάπτυξη των χωρών γειτονίας και Θέλουμε να εξασφαλιστεί ότι η επερχόμενη ε, διάσκεψη κορυφής ε, της ε, Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης του Ιουνίου θα προσφέρει νέο δυναμισμό και θα, θέσει, θα θεσπίσει νέους στόχους για το μέλλον. Η Ανατολική Εταιρική Σχέση είναι μια μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό είναι σημαντικό. Εν κατακλείδη, Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης για την υποστήριξη που προσέφερε στη δουλειά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εποχή που συνεργαζόμαστε με τους εταίρους, κυρίως στο τομέα της, του διεθνούς εμπορίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για το S&D, Ευχαριστώ λέει η κυρία Ροντρίγκεθ Πινέιρο. Ο κύριος Μιχαήλ Ντουντός δεν μπόρεσε να έρθει εδώ και έχει ετοιμάσει μία παρέμβαση. Εξ ονόματος της και Δημοκράτων θα ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν σε αυτή την ανατολική εταιρική σχέση να οδεύσει προς μεγαλύτερη ευάθυνση. Δυστυχώς η γεωγραφικές εξελίξεις ε, έχουν σοβαρό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της εταιρικής σχέσης. Θεωρώ ότι δύο βασικοί όροι προαπαιτούνται προκειμένου να υπάρξει και στο μέλλον αυτή η προνομιακή σχέση. Καταρχάς, ε, να αυξηθεί η ταχύτητα και ποιότητα των μεταρρυθμίσεων στις χώρες Ανατολικής Γενιτονίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι, δεν αποτελούν χάρη που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ένα θέμα το οποίο θα ωφελέσει τους πολίτες. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά την αύξηση της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει η υποστήριξη αυτή να μεταφράζεται σε συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα, τα οποία θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών καθημερινά. Οι πολίτε των χωρών αυτών τη Ανατολική Γειτονία έχουν ήδη επωφεληθεί από μία σειρά μέτρων, όπω η απελευθέρωση στις θεωρήσεις για τη Μολδαβία το 2014, για την Γεωργία και την Ουκρανία το 2017 και σύντομω και με τη Λευκορωσία. Η ευρωπαϊκή υποστηρίξη έχει να κάνει κυρίως ε, και με την ε, ε, Πρέτρο ανάπτυξη των υποδομών και την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων. Πολλά θα πρέπει να γίνουν ακόμα για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των πολιτών στις χώρες αυτές. Και για να πετύχουμε και μια συνεχτική και ευρεία σύνδεση. Θα πρέπει επίσης να δούμε και τη σύνδεση με τον αγωγό που μας συγγένει με την, μεταξύ Ρουμανίας και Μολδαβίας. Τα θέματα ενέργειας και ασφάλειας θα, θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο για την ευρωπαϊκή πολιτική σε ό,τι αφορά τις εταιρικέ σχέσεις στην γειτονία μας. Θα ήθελα να τονίσω παράλληλα ότι όλε αυτέ οι χώρε, εκτό από την Λευκορωσία, έχουν ε, διάφορες παγωμένες σειράξεις στην επικράτειά τους. Και όλοι ξέρουμε πώς επηρεάζουν αυτές οι τριβές το επιχειρηματικό κλίμα. Υποστηρίζω επίσης την ε, γραμμή του εισηγητή σε ό,τι αφορά την επισήμανση του θέματος της διαφθοράς και της ολιγαρχίας στην διακυβέρνηση. Θα πρέπει να καταπολεμήσει, να καταπολεμηθεί η διαφθορά και να βοηθηθούν και τα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς για να υπάρχει μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα και καλύτερος σχεδιασμός σε ό,τι αφορά το βιωτικό επίπεδο. Και σε ό,τι αφορά την, το σκέλος της συμμετοχής των ΙΠΑ αποτελούν σημαντικό στοιχείο σε ό,τι αφορά τα μακροοικονομικά ε, μέσα. Και τώρα θα ήθελα και εγώ να προσθέσω δύο πράγματα. Θα ήθελα να λάβουμε υπόψη στη γνωμοδότηση το σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των ικανοτήτων και που μπορεί να προκαλέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κοινωνία των πολιτών. Και επίσης η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει τεχνική αρρωγή στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας για να ε, ενισχυθεί το εξωτερικό πλαίσιο επενδύσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, προστασία και τη βεβαιότητα των επενδύσεων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, λέει και πρόεδρο. Από το Renew τώρα το λόγο έχει η Κάρεν. Ευχαριστώ. Και εγώ θα πάρω το λόγο ε, εξ ονόματο του κυρίου Άρμας, ο οποίο επίσης μου έδωσε τα σχόλιά του οι χώρε ανατολικής γειτονία αποτελούν βασικό σωτέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ισχύει ασφαλώ και σε ό,τι πρώτο εμπόριο. Οι έξι χώρε από κοινού αποτελούν τον δέκατο εμπορικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί βασικό εμπορικό εταίρο για την Γεωργία, την Κροατία, το Αζερβαϊτζάν, τη Μολδαβία και ο δεύτερο μεγαλύτερο για την Λευκορωσία και την Αρμενία. Είναι επίση μεγάλο δωρετή η Ευρωπαϊκή Ένωση και επενδυτή η συμφωνία εταιρική σχέση και αυτή η βαθιά συνεκτική εμπορική σχέση έχουν βελτιώσει τις σχέσεις με την ε, Μολδαβία, την Ουκρανία και τη Γεωργία και τις έχουν φέρει σε νέο επίπεδο. Η επιτυχής εφαρμογή των συμφωνιών αυτών αποτελεί κλειδί για να ακολουθήσουν περαιτέρω του ευρωπαϊκού αυτό δρόμο. Κατά πολέμηση επίσης διαφθοράς, το κρατός δικαίου. Αυτά θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό κλίμα και θα ενθαρρύνουν τι επενδύσει στην ε, περιοχή. Να τονίσω επίσης τη σημασία για μια πλατφόρμα για τη δημοκρατική ανάπτυξη και τον δημοκρατικό χώρο για την κοινωνία των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει όλη τη τεχνική και οικονομική αρρωγή για τις μεταρρυθμίσεις και για την υλοποίηση των συμφωνιών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, ευχαριστούμε τον εισηγητή. Ευχαριστώ, λέει και πρόεδρο. Δεν έχουμε κάποιον άλλον ε, σκιώδη παρόντα. Ζητά κανεί το λόγο. Το λόγο λοιπόν έχει τώρα τον κύριο, στον κύριο Βασίλη Μαραγκό. Α, δεν είναι εδώ. E Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θέλει να ξεκινήσει. Η κυρία Άννα Ευχαριστώ που μας δίνει το λόγο. Ευχαριστώ για τη συζήτηση και για την πρωτοβουλία που έλαβε αυτή η Επιτροπή σας για να συνεισφέρει στη σύσταση της ΑΦΕΤ. Είναι μια πολύ επίκαιρη συζήτηση και όπως ξέρετε πέρυσι το Συμβούλιο είπε στην Κομισιόν και στην ύπατη εκπρόσωπο να ετοιμάσει μακροπρόθεσμους ε, στόχους ε, πολιτικής για το, την περίοδο μετά το 2020. Ολοκληρώνουμε αυτή τη στιγμή μία κοινή ανακοίνωση, ένα έγγραφο δηλαδή, για να μιλήσουμε για τους μελλοντικούς ε, στόχους πολιτικής που θα υιοθετηθούν το Μάρτιο. Και συνεχεία θα ακολουθήσουν συμπεράσματα του Συμβουλίου και προετοιμασία της δήλωσης της Συνόδου Κορυφής, όπως είπατε σωστά, που θα γίνει τον Ιούνιο και μάλιστα στις 18 Ιουνίου. Τώρα, για τους μελλοντικού στόχους βασιζόμαστε στα αποτελέσματα μιας διαβούλευσης που ξεκίνησε πέρυσι. Ήταν μια πλατιά χωρίς αποκλεισμούς διαβούλευση Είχαμε πάνω από 200 συνεισφορές από συμφεροντούχους στα κράτη-μέλη, στις χώρες-μέλη, από τα θεσμικά όργανα, από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, από τις επιχειρήσεις, από τον ακαδημαϊκό χώρο, από απλούς πολίτες. Δεν θα μακρηγορήσω. Θέλω να τονίσω δύο βασικά συμπεράσματα αυτής της διαβούλευσης. Πρώτον, ότι αυτή η πολιτική γειτονίας δίνει αποτελέσματα, συγκεκριμένα αποτελέσματα, κυρίως στην οικονομία, στο εμπόριο. Τα εντυπωσιακά νούμερα ακούστηκαν από τους βουλευτές σε ό,τι αφορά την συνδεσιμότητα, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Λιγότερα εντυπωσιακά δυστυχώ είναι τα αποτελέσματα στο κράτος δικαίου και στον τομέα της ε, διακυβέρνησης, όπου πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Δεύτερο συμπέρασμα από την διαβούλευση που κρατάμε είναι ότι το τρέχον πλαίσιο το, μέχρι το 2020 οι τέσσερις πυλώνες που εντοπίστηκαν στην Ρήγα είναι σωστοί και εξακολουθούν να ισχύουν όπως και η αρχιτεκτονική, η δομή το, που έχουμε θεσπίσει για τη συνεργασία και διμερός αλλά και πολυμερός. Προτεραιότητες. Προφανώς, πολλές από τις συνεισφορές που λάβαμε βάλαν την οικονομία ως πρώτη προτεραιότητα. Ανάπτυξη, θέση απασχόληση δηλαδή. Είναι η πρώτη ανησυχία, το πρώτο μέλημα και η βασική προτεραιότητα για τη συνεργασία με τις χώρες αυτές. Και πολύ σωστό, όπως είπατε, υπάρχει το θέμα της ε, καταπολέμησης διαφθοράς και της διατήρησης του κράτους δικαίου. Βασική προϋπόθεση για οτιδήποτε άλλο. Και για να κλείσω, επιβεβαιώνω ότι και οι συνεισφορές και η μελλοντική πολιτική θα επιμένουν στην ανάγκη πλήρους ε, εφαρμογής ε, των συμφωνιών σύνδεσης και των ε, συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου και αυτό θα παραμείνει βασική προτεραιότητα και στο μέλλον. Θα σταματήσω εδώ. Περιμένω και να γίνουν και περαιτέρω συζητήσεις εν ώψη της Συνόδου Κορυφής και πριν τη Συνόδου Κορυφής. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Καλημέρα. Ε, εκ μέρους της ε, Γενικής Διεύθυνσης ΝΙΑΡ Καλημέρα σας. Ακούσατε τα σχέδια για τη νέα ανακοίνωση πριν από λίγο. Ε, ετοιμάζουμε μαζί με τις υπηρεσίες και τα κράτη-μέλη το κείμενο αυτό και ελπίζουμε ως ονούπο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να διατηρήσουμε μαζί την ενότητα και τη συνένεση που υπάρχει για αυτή την αρκετά επιτυχημένη πολιτική, όπως όλοι ξέρουμε. Και όπως αποδείχτηκε στις διαρθρωμένες διαβουλεύσεις που ξεκίνησαν στα πλαίσια της 10ης ε, επαιτίου. Αυτό που προέκυψε από τις διαρθρωμένες διαβουλεύσεις είναι μια αναγνώριση ότι το πλαίσιο, το συνολικό πλαίσιο ε, για το χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2020 έδωσαν αυτά αποτελέσματα για την κοινωνία των πολιτών, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, αλλά και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις δρομολογήθηκαν ε, και τις υποδέχτηκε ο κόσμος θετικά και θεωρείται λοιπόν πολύ καλό το πλαίσιο αυτό και για το μέλλον. Να δώσω δύο-τρία σχόλια ακόμα για το μέλλον και τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών και πώς εφαρμόζουμε τις συμφωνίες σύνδεσης αλλά και τις υπόλοιπες συμφωνίες που έχουμε με τις χώρες της περιοχής. Στο παρελθόν, μαζί με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου μετασχηματίσαμε, αλλάξαμε τις σχέσεις που έχουμε με την κοινωνία των πολιτών, αλλά και με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Γιατί πολύ, πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι ε, της βοήθειάς μας περνάει μέσα από την ανάμιξη των χρηματοδοτικών μέσων, το blending, για να υπάρχει ε, επίδραση στην πραγματική οικονομία. Και αυτό ήταν ε, πολύ σημαντικό στο παρελθόν. Στο πλαίσιο των βαθιών και σφαιρικών αυτών ε, συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου έχουμε αυτές τις, αυτούς τους μηχανισμούς ε, με τις τρεις χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία και τώρα ε, για την συμφωνία με την Αρμενία ε, έχουμε επεκτείνει την υποστήριξη και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αρμενίας. Και σκεφτόμαστε πώς θα το αναπτύξουμε περαιτέρω και στις άλλες δύο χώρες που συμμετέχουν στην ανατολική εταιρική σχέση. Σε ό,τι αφορά την κοινωνία των πολιτών, έχουμε συμφωνίες εταιρικής σχέσης με μεγάλες οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών κυρίως, αλλά και έχουμε προχωρήσει από την εφαρμογή των σχεδίων από την κοινωνία των πολιτών στην εμπλοκή, στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή οι ακτιβιστές οι ίδιοι, τα μέλη ας πούμε των οργανώσεων λοιπά συμμετέχουν για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για καλύτερες ε, υπηρεσίες στους πολίτες. Επομένως η κοινωνία των πολιτών είναι φορέας, είναι υπεύθυνη όχι μόνο για τις μεταρρυθμίσεις, αλλά γιατί γεφυρώνει το χάσμα ε, ανάμεσα στους πολίτες και στο πολιτικό επίπεδο, στους φορείς. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις συνεισφορές κατά τις διαρθωμένες διαβουλεύσεις και να προτείνουμε μία νέα φιλοδοξία υπογραμμισμένη. Ένα νέο φιλόδοξο πλαίσιο που θα συνεισφέρει στη σταθερότητα, ασφάλεια, ευημερία της ανατολικής γειτονία μας να είναι ανθεκτικές αυτές οι χώρες. Ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία της παγκόσμιας στρατηγικής μας, ειδικά σε ό,τι αφορά τη γειτονία. Τονίζουμε ακόμη περισσότερο την ανθεκτικότητα, την αντοχή, κυρίως ανθεκτική οικονομία, κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικές, αλλά και ανθεκτικοί φορείς, κράτος δικαίου και τελευταίως περιβάλλον. Περιβάλλον και κλίμα που να αντέχει. Αυτό το συζητήσαμε τις χώρες εταίρους και περιμένουμε ότι θα θελήσουν να εμπλακούν σε μια νέα προσαρμοσμένη εκδοχή της Πράσινης Συμφωνίας ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική αντοχή, βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των χωρών και προσαρμοσμένες στις χώρες. Επίσης, θα εστιάσουμε στη στρατηγική επικοινωνία. Το έχουμε κάνει ε, στο παρελθόν μέσω ε, ενός εμπορικού σήματος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε το EU for Business, Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Επιχειρήσεις, που είναι ένα πλαίσιο για όλες τις δραστηριότητες που υποστηρίζουν τον ιδιωτικό τομέα. Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ενέργεια, για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Γεωργία, Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αρμενία. Βασιζόμαστε όμως αυτό και θα δουλέψουμε ακόμα πιο στενά με όλους τους εταίρους το κάναμε με τα κράτη-μέλη, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε περισσότερο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να φέρουμε στους πολίτες και σε τοπικό επίπεδο τις πληροφορίες για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι τους προσφέρει. Μια τελική κουβέντα για την διαφοροποίηση και την ένταξη. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, μαζί με την ευελιξία και την εστίαση της αναθεωρημένης πολιτικής για την Ανατολική Γειτονία ήταν ψηλά στις ε, προτεραιότητες των ε, ομιλητών στη διαβούλευση αυτή που κάναμε. Ε, θέλουμε μια καλύτερη διαφοροποίηση ανάμεσα, ε, ισορροπία συγγνώμη, ανάμεσα στη διαφοροποίηση και στην ένταξη, γιατί όλες οι χώρες είναι διαφορετικές. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένταξη χωρίς αποκλεισμούς. Οι χώρες θα πρέπει να ανταλλάσσουν, να συνομιλούν με εμά και μεταξύ τους και θα πρέπει όμως να τις μεταχειριστούμε διαφορετικά, γιατί έχουν άλλη φιλοδοξία και άλλο ρυθμό μεταρρυθμίσεων η μία από την άλλη. Η διαφοροποίηση λοιπόν ε, λαμβάνεται υπόψη κυρίως σε διμερές επίπεδο, όπως ξέρετε, και η αντολική εταιρική σχέση, περιμένουμε, και αυτό θα είναι θύμα των προτάσεών μας, θα παραμείνει ευέλικτη και στοχευμένη στα συμφέροντα, τη φιλοδοξία και την πρόοδο που σημειώνει ο, ο κάθε ε, τέρος. Και το more for more, ε, περισσότερα θα κάνουμε εμείς όταν κάνουν περισσότερα οι χώρε. Δηλαδή αυτές οι χώρε που κάνουν περισσότερες μεταρρυθμίσει, εμείς θα, τις, θα το λαμβάνουμε υπόψη μα και θα, τις, ε, θα έχουμε μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με αυτέ. Θα βασιστούμε λοιπόν στη δουλειά που κάναμε στο παρελθόν, αλλά δεδομένων των σημερινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε την Πράσινη Συμφωνία, στον ψηφιακό τομέα, μια το χτίσιμο μιας ε, κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, μπορούμε λοιπόν να έχουμε περισσότερες επαφές με τους εταίρους που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ, η συγγήτρια. Δεν έχω περαιτέρω σχόλια. Ευχαριστώ. Η 24 Φεβρουαρίου, τελική προθεσμή υποβολής τροπολογιών, στις 12 το μεσημέρι. Και η Ψηφοφορία στις 16 Μαρτίου. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 9. Επίσης, ε, σύσταση της ΑΦΕΤ για τα θέματα των Δυτικών Βαλκανίων. Επίσης, ένα ενδιαφέρον θέμα. Ο κύριος Μπουτικόφερ είναι ο συντάκτης γνωμοδότησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως όλοι γνωρίζετε αρκετά καλά, υπάρχει πάρα πολύ περιορισμένος χώρος για γνωμοδότηση πάντα έτσι έχω περιοριστεί στα 10 σημεία, τα, οποία, τα περισσότερα εκ των οποίων θα τα βρείτε απολύτως ξεκάθαρα. Αλλά υπάρχουν και αυτά που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν, να προκαλέσουν κάποια συζήτηση. Είναι το 4 που ασχολείται με την ε, FTA της οικονομικής ε, ε, Ένωσης Ευρασίας με την ε, και όχι. Ε, το 6 είναι πολύ προσεκτικά, επιφυλακτικά διατυπωμένο, επισημαίνει την ανάγκη καλών σχέσεων γειτονίας, ασχολείται με μια από τις βασικές συγκρούσεις, συγκεκριμένα αυτή της Σερβίας με το Κοσφοπέδιο, ε, το σημείο 7 επικεντρώνεται στην ανάγκη όπως θεωρώ εγώ, να δοθεί υψηλή προτεραιότητα ε, στην περιοχή αυτή στο πλαίσιο της στρατηγικής συνδεσιμότητας της Ένωσης. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για συνδεσιμότητα αν δεν κινηθούμε στην άμεση γειτονιά μας και τα τελευταία δύο σημεία ασχολούνται με τη διάσταση της ενέργειας και υπογραμμίζουν την ε, ανάγκη να επιμείνουμε σε προγράμματα που συνάδουν με τους ε, κλιματικούς στόχους στην περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, όπως επίσης και τις διατάξεις της ε, συνθήκης για την ενεργειακή κοινότητα. Και τώρα η κυρία Γκιώρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω ουγγρικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του. Ξεκίνησαν όλα με μια δυσκολία. Η έκθεση έπρεπε να είναι έτοιμη πριν δημοσιεύσει η, τη στρατηγική της διεύνησης η παρούσα επιτροπή, δηλαδή στις 5 Φεβρουαρίου. Γι' αυτό προτείνω να ενσωματώσουμε τα κομμάτια περί εμπορίου στο έγγραφο αυτό. Θα ήθελα να υπάρξει αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον, ε, και τον όρο της αμοιβαίας εμπιστοσύνη στην έκθεση, όπως επίσης και μια ε, αμοιβαία προσέγγιση. Τώρα, το Κοινοβούλιο και ο εισηγητής είναι υπέρ της διεύρυνσης. Οι εταίροι είναι σημαντικοί σημαντικότατη εταίρη της Ένωσης και το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου τους ε, κατευθύνεται προς την Ένωση 67% των εισαγωγών και 80% των εξαγωγών τους ε, κινούνται προς και από την Ένωση. Πρέπει να δούμε ότι από το ε, ωφελούμεθα. 9 δις ευρώ είναι το εμπορικό πλεόνασμα της Ένωσης. Εάν ε, δείτε τη συνολική εικόνα, διαπιστώνετε ότι η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων έχει προσαρμοστεί σε εμά. Όμως εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε πότε θα υλοποιηθεί η διεύρυνση. Δείτε το σημείο 4, το οποίο αναφέρει ότι ανησυχεί για τις δράσεις της Σερβίας εγώ θα ήμουν προσεκτική. Δεν θα ήθελα να ε, κατονομάζω κάποιους. Ε, δηλαδή θα άλλαζα τη διατύπωση λέγοντας ότι ζητάμε από τις υποψήφιες χώρες να όταν αναπτύσσουν εμπορικές πολιτικές να λαμβάνουν υπόψη τη μελλοντική ένταξή τους στην Ένωση ώστε αυτή να συνάδει με τις εμπορικές πολιτικές της Ένωσης. Πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για κυρίαρχα κράτη. Έχουμε ήδη, τους έχουμε ήδη επιβάλει πολλά στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της ε, διεύρυνσης. Του αναμένουμε από αυτούς να έχουν συγκεκριμένες επιδόσεις και να τηρήσουν αυστηρές απαιτήσεις που είναι δύσκολο να τηρηθούν. Εγώ θα ήμουν πιο ήπια όσον αφορά το σημείο 4. Μετά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα να ε, εμφανίζονται περισσότερο στο κείμενο. Και επίσης, κάτι άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει την Σερβία και την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την ένταξή τους στον ΠΟΕ. Οι άλλες τρεις χώρες είναι ήδη μέλη του ΠΟΕ. Πρέπει και αυτές να γίνουν. Ευχαριστώ. Thanks a lot. Ευχαριστώ όλοι και πρόεδρος για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες στο λογοχήμα. Εδώ είμαι και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μιλάω εξ ονόματος του κ. Μπέικερ, ο οποίος δυστυχώς επίσης δεν ε, μπορεί να παρευρεθεί. Η στρατηγική λοιπόν αυτή είναι στρατηγική σημασία για την ε, ε Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι διεύρυνση. Επιτρέπει λοιπόν ένα σαφέ ε, μονοπάτι για την ανάπτυξη για τις χώρες αυτές σε ό,τι αφορά και τις φιλοδοξίες τους και ό,τι αφορά το εμπόριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και προς την με, πριν από το 2020 για τα Δυτικά Βαλκάνια, θα πρέπει να επιβεβαιώσει την δεσμευσή μα σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει μα με τη Σερβία και το Μαυροβουνίο, την ακίνηση των διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και την διευκόλυνση ενό ε, σαφού, σαφούς δρόμου προ την διευρύνση, προ την ένταξη για τι υπόλοιπε χώρε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό δεδομένο και των καθυστερήσεων των τελευταίων χρόνων σε ό,τι αφορά την εκκίνηση διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία. Η σύστασή μα λοιπόν θα πρέπει να λάβει υπόψη τη νέα μεθοδολογία για τι διαπραγματεύσει για την προσχώρηση που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα δώσουν σαφεί κατευθυντήριε γραμμέ και θα δώσουν δυνατότητα να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει για κεφάλαια τα οποία έχουν ήδη κλείσει όταν δεν έχουν ε, διαπιστωθεί πραγματικά η εκτέλεση των μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει να, καλώς, να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε τις χώρες για τις μεταρρυθμίσεις αυτές σε ό,τι αφορά τα θεσμικά όργανα, το κράτος δικαίου και ένα οικονομικό σύστημα με ίσους όρους για όλους τους ε, παράγοντες. Να μπουν κλείδες ασφαλείας για την προστασία των επενδυτών, έγκριση των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εργασιακά και τα κοινωνικά δικαιώματα. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες είναι σημαντικό η προσχώρηση σε ό,τι αφορά τα Βαλκάνια να μην συμβάλλει μόνο στην ανταγωνιστικότητα και στο εμπόριο. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε και την ευημερία, τα πρότυπα διαβίωση, τι προοπτικέ και τη γενική ε, κοινωνική ευημερία. Είναι σημαντικό να συνεχίσει η οικονομική συνεργασία για να υπάρξει διαφορετική συνδεσιμότητα και να υπάρξει υπεραιτέρω ανάπτυξη του χώρου εμπορίου. Να καλέσουμε εμείς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνουν μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική αρρωγή σε ό,τι αφορά το εργαλείο για την πρωτεξιακή βοήθεια. Να τονίσω επίσης ότι πιστεύουμε ότι ο εισηγητής έκανε πολύ καλή δουλειά και θα συνεργαστούμε στενά για να λάβουμε υπόψη όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέραμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και για το Renew τώρα. Η κυρία Τσάντσοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Καράντσοβα. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί εκτιμώ τη θετικό τόνο που έχει. Είναι σημαντικό αυτό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα τα θετικά μηνύματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τονίζουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τις χώρες αυτές. Θέλουμε να στείλουμε και ένα μήνυμα επιπλέον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση και είναι έτοιμη να δώσει πιο πολύ πνοή σε αυτή τη διαδικασία. Να δούμε επίσης πώς μπορούμε συγκεκριμένα να υποστηρίξουμε τις χώρες αυτές πώς μπορούμε να τις κάνουμε να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από τις συστάσεις που ήδη περιλαμβάνονται. Θα ήθελα να τονίσω και κάποιους άλλους τομείς που θα πρέπει να αναφέρουμε. Να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε έργα από το Ταμείο για τα Δυτικά Βαλκάνια και να υποστηρίξουμε το εργαλείο για την προτεξική βοήθεια. Τομείς προτεραιότητας ιδιαίτερα για τις ε, εμπορικές μας σχέσεις είναι υποδομές ε, για τις ε, μεταφορές που είναι σημαντικό στοιχείο για τις συναλλαγές με την περιοχή αλλά και για να σταθεροποιήσουν το επιχειρηματικό κλίμα. Θα πρέπει να προωθήσουμε επίσης τις περιφερειακές ρυθμίσεις Schengen ως ένα βήμα για την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανοίγοντα σιγά σιγά τα σύνορα να προετοιμαστούν οι χώρε για την ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλο, εδώ στην γραμματότηση να τονίσουμε και κάτι που είπαν οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει ενεργά να υποστηρίζει τι συζητήσει για την προσχώρηση στον ΠΟΕΔ με τη Βοσνία και τη Σερβία. Αυτά λοιπόν θα ήθελα να προσθεθούν στην γνωμοδότηση και σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Εσιάρ, ο κύριο Σάρντι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, η χώρα μου υποστήριξε παραδοσιακά οποιαδήποτε διεύρυνση της Ένωσης. Πιστεύω σε εκ τούτου ότι εμείς στην Ένωση πρέπει να είμαστε σαφείς στις ενδείξεις που δίνουμε για την προοπτική ένταξη στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Από την άλλη πρέπει να πω ότι έχω και κατανόηση για τα κράτη-μέλη που αισθάνονται ε, την ε, κόποση της διεύρυνσης και μπορώ να ε, αντιληφθώ για ποιο λόγο υφίσταται αυτό το φαινόμενο. Άρα πρέπει να επιμείνουμε να ε, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δεσμεύσεις πριν από οποιαδήποτε ένταξη. Όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης, ε, τη θεωρώ ευπρόσδεκτη. Συμφωνώ με τα βασικά πολιτικά μηνύματά της. Δύο σημεία μόνο Πρώτον, πιστεύω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε πιο, με μεγαλύτερη έμφαση ε, την ε, ανάγκη αντιμετώπισης της διαφθοράς και την ανάγκη για ε, χρηστή διακυβέρνηση. Γνωρίζουμε ότι οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στους τομείς της χρηστής διακυβέρνησης και της διαφθοράς. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αποφεύγουμε να πούμε ακριβώς τι παρατηρούμε και να επιμείνουμε να βελτιωθεί η κατάσταση στο άμεσο μέλλον. Όσον αφορά την ενέργεια, πρέπει να ληφθεί υπόψη ένα θέμα σημαντικό. Ήτι, ε, ε, υπάρχει έλλειψη παροχής ενέργειας στην περιοχή και το πιο σημαντικό στοιχείο για τις χώρες αυτές είναι να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια όπως ονομάζουμε ε, στην περιοχή είναι σημαντικό ο τομέας της ενέργειας να καθοδηγήσει ε, της, ε, την οικονομική ανάπτυξη μέσω ε, πολυμερών συνεργασιών σε έργα όπως ο, ο βόρειος άξονας φυσικού αερίου. Κατά τα άλλα νομίζω ότι είναι καλά τα πράγματα και θα υπάρξει στο τέλος θετικό αποτέλεσμα. Αν δεν υπάρξει ε, άλλος που θέλει να πάρει το λόγο, δίνω το λόγο στην Επιτροπή, στην τον κύριο Κοβάλσκι. Α, όχι, κάποιος άλλος θέλει τον, ε, τον λόγο. Συγγνώμη. Δύο λόγια μόνο. Είναι σχέδιο γνωμοδότησης που περιλαμβάνει πολύ περισσότερες ε, πτυχές από η έκθεση της ΑΦΕΤ. Ε, υπάρχει και πρόκληση ε, κάπου, δηλαδή ε, Υπάρχει το θέμα της ενισχυμένης, ε, αναλογι... Ε, ενισχυμένης αναλογίας. Παρά τα αυτά, το, το κείμενο είναι σωστό. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε για αυτή καθεαυτή τη διεύρυνση. Αν το μόνο σχέδιο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι μια διεύρυνση χωρίς όρια, χωρίς αμφισβήτηση, μια ατελείωτη διεύρυνση, κάποιες χώρες, συγκεκριμένα η δική μου, ε, η Γαλλία, θα έχουν προβλήματα προβλήματα, προβλήματα συνεννόησης μεταξύ μας. Γιατί αν η Ευρώπη είναι απλό και μόνο μια μεγάλη αγορά, να συνεχίσουμε τη διεύρυνση χωρίς όρια. Αν όμως αντιστοιχεί σε ένα πολιτικό ε, σε μια, πολιτική, σε μια πολιτική προσπάθεια, τότε υπάρχουν πολλές χώρες και εγώ ως ε, τη δική μου χώρα τη γνωρίζω που είναι και ιδρυτική χώρα ε, πιστεύω ότι θα υπάρξουν άγχοι ερωτηματικά που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει φόβος να καταστραφεί όλο το οικοδόμημα. Με τα φυσικά τα Βαλκάνια, η, η σχέση μας με τα Βαλκάνια είναι πολύ σημαντική. Αλλά αν πρέπει να επισπευθεί η διαδικασία διεύρυνσης ε, χωρίς ε, όρια, αυτό δεν Γι' αυτό δεν είμαι βέβαιος. Ευχαριστώ. Και τώρα, και τώρα ο κύριος Κουβάλσκι. Καλημέρα σας. Δύο λόγια για την προσέγγιση της Επιτροπής και την δουλειά που κάνει η Επιτροπή στην περιοχή αυτή. Έγινε το, πρώτο εξάμεινο που που συνεχίζει το έργο τη, των πολλών προηγουμένων ετών. Επικεντρωνόμαστε σε τρία ζητήματα. Αναφερθήκατε στην ανακοίνωση για την αναθεωρημένη μεθοδολογία της διεύρυνσης της αρχής Φεβρουαρίου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ε, πρόοδος στην άνοιγμα των διαπραγματεύσεων με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και επίσης είναι ευπρόσδεκτη η ε, και δουλεύουμε για ε, μια ανακοίνωση επιτροπής για ένα ε, ουσιαστικό σχέδιο οικονομικών επενδύσεων στην περιοχή που προσβλέπουμε να παρουσιαστεί το Μάιο στο Ζάγκρεπ. Τώρα, το σχέδιο αυτό οικονομικών επενδύσεων θα δώσει μεγάλη έμφαση όχι μόνο στις οικονομικές επενδύσεις και στην στήριξη των οικονομικών παραγόντων, αλλά θα δώσει έμφαση στο κράτος δικαίου και θα υπάρξει και μια σημαντική ε, πράσινη ε, ε, διάσταση που αναφέρθηκε ρητά στην ε, ανακοίνωση της Κομισιόν για το Green Deal. αυτό, αυτή η γνωμοδότηση είναι ευπρόσδεκτη. Η περιφερειακή συνεργασία, η περιφερειακή συνεργασία αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της επιτυχίας αυτού του σχεδίου. Ενδεχομένως θα είδατε ή θα έχετε διαβάσει ότι υπάρχει μια μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας που επισημαίνει ότι η ευρύτερη και βαθύτερη ολοκλήρωση της αγοράς στα Δυτικά Βαλκάνια μπορεί να οδηγήσει ε, σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 6,7 ε, μονάδες. Πράγμα πολύ σημαντικό. Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με την περιοχή μέσω της περιφερειακής οικονομικής περιοχής, τέσσερις πυλώνες, εμπόριο, επενδύσεις, κινητικότητα και το ψηφιακό θεματολόγιο. Το θεματολόγιο που είναι ουσιαστικά το πολιετές πρόγραμμα δράσης στην Τριέστη, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του 2017 ο χώρος ελευθέρου εμπορίου στηρίχθηκε στο ΣΕΦΤΑ. Έχουν γίνει πρόοδοι εδώ με κάποιες συμφωνίες που τελικά συνήφθησαν. Η, το πολιετές σχέδιο της περιφερειακής οικονομικής, του περιφερειακού οικονομικού χώρου επικεντρώνεται στην δημιουργία ενός δημιουργία κοινών επενδυτικών προτύπων, ώστε οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων να τα χρησιμοποιήσουν κατά την ε, διαπραγμάτευση των διμερών επενδυτικών συμφωνιών τους για να μπορούν να ευθυγραμμιστούν με τις βέλτιστες πρακτικές της Ένωσης στον τομέα αυτό. Έχει σημειωθεί πρόοδος εκεί. Επίσης, συνεχίζουμε την υποστήριξή μας προς τον ιδιωτικό τομέα της περιοχής. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε συνεισφέρει σε περιφερειακά εργαλεία για πρόσβαση στην, τα, ε, ε, σε χρηματοδότηση είναι πάνω από 320 εκατομμύρια ευρώ που έχει δημιουργήσει ε, ιδιωτικό κεφάλαιο επενδύσεων πάνω από 3,7 δις ευρώ και το ενδιαφέρον μας για την περιοχή ήταν και ένα ε, εργαλείο εγγυήσεων των επενδύσεων 150 ε, εκατομμυρίων που πιστεύουμε ότι θα μοχλεύσει την αρχική αξία του κατά 10 φορές. Αρχικά προς... θέλουμε να διευρύνουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Βιώσιμων Επενδύσεων στα Δυτικά Βαλκάνια για τη στήριξη των επενδύσεων. Θα υπάρξει σημαντική συνέχιση του έργου συνδεσιμότητας στη νέα ανακοίνωση που ετοιμάζουμε ενώπιση του Ζάγκρεμπ από το 2014 μέσω του πλαισίου επενδύσεων ε, Δυτικών Βαλκανίων έχουμε ένα έργο 880 εκατομμυρίων ευρώ που έχει μοχλευθεί σε 2,3 δις με ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό για βασικά έργα συνδεσιμότητας, οδικές μεταφορές και σιδηροδρομικές μεταφορές και έργα ενεργειακά. Και αυτά θα συνεχιστούν και θα ενταχθούν στην ε, νέα ανακοίνωση. Τέλος, όσον αφορά την πράσινη ατζέντα, προτείνουμε να σκεφτούμε και να φανούν εκεί τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Green Deal ως το δυνατόν περισσότερο, αλλά τα οποία θα προσαρμοστούν στην πραγματικότητα ε, επιτόπου. Ευχαριστώ. Τέλεια. Αυτό το Green Deal είναι ένα είδος ε, κάτι που υπάρχει παντού, αλλά δεν είναι συγκεκριμένο, είναι λίγο μυστήριο. Πρέπει φυσικά να σκεφτούμε ώστε να γίνει αυτή η εταιρική σχέση πιο πράσινη. Yes, uh, Mr. Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης, ο κ. Ράμπερτ. Καλημέρα. Οι συνάδελφοι της Κομισιόν έφεραν διάφορα πράγματα, τα οποία δεν θα επαναλάβω. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία ε, για να φτιάξουμε ένα πλαίσιο για κάποιες από τις προτάσεις ε, που έχει κάνει η ΙΝΤΑ για να και προτάσεις δηλαδή ενσωμάτωση, ενσωμάτωση στο... στην πρόταση ψηφίσματος. Σημειώνω ένα-δύο πράγματα που ανέφερε και η Κομισιόν και τα υπογραμμίζω για... και που είναι σημαντικά και για την την, ε, τον υπατοεκπρόσωπο. Ε, συμφωνούμε με την, ε, τις διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία και ελπίζουμε να βρεθεί συνένεση για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τις δύο αυτές χώρες, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία. Επίσης, ε, τονίζουμε ότι η αναθεωρημένη μεθοδολογία της Κομισιόν λαμβάνει υπόψη όλες τις διαφορετικές θέσεις στο Συμβούλιο και αντικατοπτρίζει σωστά το σημείο ισορροπίας και Πιστεύουμε ότι ο εξυγχρονισμός της διαδικασίας διεύρυνση και η, η έναξη ενταξιακών, διαπραγματεύσεων θα πρέπει να γίνουν από κοινού. Θα ήθελα να σταθώ στο σημείο 4 των προτάσεων σε ό,τι αφορά την ε, ε, υπογραφή συμφωνίας ε, με τη Σερβία. Έχουμε κοινέ ανησυχίες για την επιρροή τρίτων χωρών στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Η Σερβία μπορεί να κάνει συμφωνίες με άλλες χώρες πριν από την ένταξη της Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να σέβεται τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Σερβία υπό την Συμφωνία Σταθεροποίηση και Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση Σερβία και κάθε φορά θα αξιολογούμε τι ε, υποθέσει αυτέ αναπερίπτωση. ό,τι αφορά τι ε, πρωταξιακέ διαπραγματεύσει, η Σερβία έχει ε, δεσμευτεί να αποσυρθεί την ημέρα τη ένταξή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από όλε τι διμερεί συμφωνίε, από τι εμπορικέ συμφωνίε με τρίτε χώρε. Είναι γενικό κανόνα που αφορά όλε τι υποψηφίε χώρε που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, αξίζει να αναφέρουμε ότι η πραγματική οικονομική και εμπορική επίπτωση είναι, της συμφωνίας αυτής είναι πολύ περιορισμένη σε σχέση με τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες που έχει αυτή τη στιγμή ήδη η Σερβία. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε το μέγεθος της, του εμπορίου που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Σερβία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει το 63% του εμπορίου, του συνολικού εμπορίου με τη Σερβία το εμπόριο τη Σερβία με τη Ρωσία είναι λιγότερο το 10% του συνολικού εμπορικού όγκου τη Σερβία. Οι επενδύσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Σερβία είναι δεκαπλάσιε από τη Ρωσία. Θα ήθελα λοιπόν να τα πω αυτά εν είδη πλαισίου για να ξέρουμε τι λέμε. Οι συνάδελφοι τη Κομισιόν μίλησαν με λεπτομέρειε για τη σημασία τη ε, συνδεσιμότητα και τη περιφερειακή διάσταση που αναφέρεται στο σημείο 7 από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Για μας σημαντικό είναι και η συνδεσιμότητα και η περιφερειακή συνεργασία για την ε, περιφερειακή σταθερότητα. Είναι σημαντικό στοιχείο για να επιληθούν διμερεί θέματα μεταξύ των εταίρων το, στα Δυτικά Βαλκάνια και γενικότερα συνεισφέρουν σε ένα κλίμα αμοιβαίας συνεργασίας. Σημείο 10. Η πρόταση προσθήκης γίνεται η ανάγκη ε, τα μέλη των Δυτικών Βαλκανίων που είναι και μέλη της ενεργειακής κοινότητας να σέβονται τις διατάξεις της ενεργειακής κοινότητας αμελητή. Να σεβαστούν μάλλον αμελητή τις διατάξεις αυτές. Η προϋπόθεση ποια είναι, ότι η Σερβία θα ικανοποιήσει την Σέρβα Γκάς και την ε, Ιούγκαρος Μπάς και θα υπάρξει ανταγωνισμός και θα ε, σεβαστεί, με τη, σεβαστεί τις προϋποθέσεις της γραμματείας ενεργειακής κοινότητας και ειδικά ε, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά ε, αερίου και οι νέοι φορείς θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά. Τον Ιούνιο ε, του 19 υπήρχαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που τονίζουν την ανάγκη η Σερβία να ευθυγραμμίσει την ενεργειακή της πολιτική με το, νοσιακό και εκτιμένο ειδικά σε ό,τι αγορά την αγορά ε, αερίου και τα project, τα προγράμματα του Γκαστράν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπεντικόφερος, η μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα πολύ χρήσιμα στοιχεία τα οποία επισημαίνουν. Προσβλέπω στις τροπολογίες σας. Και σκοπεύω και εγώ να καταθέσω κάποιες τροπολογίες για κάποιες επιπρόσθετες ιδέες οι οποίες δεν χώρεσαν στο αρχικό κείμενο. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι προς την ίδια κατεύθυνση κινούμαστε. Ένα ενδεχομένως αμφιλεγόμενο θέμα είναι για το σημείο 4 για το σερφικό αυτό ζήτημα και το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να γίνει μια σωστή συζήτηση για το πόσο ανοιχτά και ειλικρινά θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Να ευχαριστήσω όλους σας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος μία η κατάθεση τροπολογιών είναι 24 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Ευχαριστώ. Τώρα να πάμε στο σημείο 10. Έκθεση GSP. Για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Πολύ σημαντικό σημείο για την εμερινή μας ατζέντα. 71 χώρες ωφελούνται άλλωστε από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Πολλές εξ αυτών βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και χρειάζονται υποστήριξη. Και φυσικά Έχουμε και κάποιες χώρες όπου θα θέλαμε να υπάρξει αξιολόγηση των δεσμεύσεών τους σε ό,τι αφορά το GSP+. Γι' αυτό και έχουμε κάποια συγκεκριμένα έγγραφα για την ε, Καμπότζα, τη Μιαμάρ και τον Μπαγκλαντές. Αυτό λοιπόν το σημείο στην ημερήσια διάταξη έχει να κάνει με το που βρισκόμαστε εν ώψη και της μελλοντικής μεταρρύθμισης του καθεστώτος του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Νομίζω ότι το 2021 αναμένεται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί το τρέχον σύστημα θα εκπνεύσει το 2023. Και αυτό λοιπόν θα κληθούμε να το συζητήσουμε ο εξυγχρονισμός του GSP και του σχετικού κανονισμού. Έχουμε μαζί μας εκπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα σας δώσω 15 λεπτά και στους δύο μαζί. Θα χρειαστεί λοιπόν να μοιραστείτε το χρόνο αυτό όπως το επιθυμείτε. επικεφαλής λοιπόν του εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης του συστήματος GSP, η κυρία Άρινα Μπότσουκ. Καλημέρα κύριε βουλευτές, κύριε βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ σήμερα για να ανταλλάξουμε απόψεις σε ό,τι αφορά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Σύστημα Γενικευμένων μόνο. Είναι η τρίτη έκδοση, η τρίτη φορά που έχουμε κάνει τη σχετική έκθεση στα πλαίσια του, του κανονισμού αυτού. Δημοσιεύτηκε και διαβιβάστηκε παράλληλα προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στις 10 Φεβρουαρίου. Η έκθεση όντω καλύπτει τις εξελίξεις σε 71 χώρες που ωφελούνται από το σύστημα αυτό και επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα στο, στις νέες χώρες GSP Plus και στις τρεις χώρες με, μέσω της ε, βελτιωμένης ε, συμμετοχής ε, στο σύστημα Anything But Arms, όλα εκτός από όπλα. Τα βασικά μηνύματα που προσπαθούμε να περάσουμε μέσω την έκθεση αυτή είναι τα εξή. Καταρχάς να αναφερθούμε στο οικονομικό σκέλος. Το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ε, υποστήριξε σωστά την ενσωματώση των χωρών αυτών στο διεθνές εμπόριο. Τα οικονομικά λοιπόν στοιχεία είναι, μιλούν για μια μεγάλη επιτυχία. Και κατά καταδεικνύουν το 2017 και 2018 οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 71 αυτές χώρες αυξήθηκαν και αγγίζουν πλέον τα 184 δις. 70 δις εξ αυτών καταχωρίστηκαν στο σύστημα GSP σε αριθμούς ρεκόρ. Έχουν αυξηθεί λοιπόν οι δικαιούχοι. 71 πλέον. Μάλλον έχουν μειωθεί οι δικαιούχοι, αλλά έχουν αυξηθεί ο όγκος των συναλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι ωφελούνται σημαντικά αυτές οι χώρες από τις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οικονομικά στοιχεία είναι πολύ ε, σημαντικά για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Στατιστικά φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις χώρες αυτές εισάγει πάνω από το διπλό όγκο από αυτό που εξάγουν αυτές οι χώρες στον υπόλοιπο κόσμο. Πρόκειται λοιπόν ένα πολύ γενναδρό σύστημα προς τις χώρες αυτές, τις οποίες και το, οι οποίες και το χρησιμοποιούν εκτενώς. Ένα άλλο στοιχείο. Κάποιες ε, χώρες έχουν ε, αναπτυχθεί αρκετά και έχουν φύγει από το σύστημα αυτό. 11 χώρες έχουν βγει λοιπόν από το σύστημα και υπολογίζουμε ότι θα μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των δικαιούχων χωρών. Βλέπουμε ότι πρόκειται και για ένα στοιχείο επιτυχίας γιατί υποστηρίζεται η οικονομική ενσωμάτωση Έχουμε φτάσει λοιπόν αυτές οι χώρες στο ανώτατο μέσο εισόδημα. Μόλις φτάνουν λοιπόν αυτό το όριο το οποίο το ορίζει η, η Παγκόσμια Τράπεζα αφαιρούνται αυτόματα από το σύστημα. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο προβάλλεται ιδιαίτερα στην έκθεσή μας είναι η συνεισφορά σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη από το πρόγραμμα, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Μιλάμε λοιπόν για την ε, ε, επικύρωση 27 συμβάσεων για το περιβάλλον, τα κοινωνικά, το εργασιακά κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο κοινωνικό διάλογο και από τα, αποτελέσματα, από τα συζητήσεις που κάνουμε από τις χώρες αυτές ότι υπάρχουν αποτελέσματα για, σε ό,τι αφορά παράδειγμα την παιδική εργασία. Να σας πούμε ότι η Σρι Λάνκα έχει εισάγει μια ζώνη χωρίς παιδική εργασία και κατάφερε να μειώσει σε εθνικό επίπεδο την παιδική εργασία σε 1% το 16% και επίσης μέχρι το 2022 έχει δεσμευτεί να καταργήσει εντελώς την παιδική εργασία και την Βολιβία να αναφέρω. Χάρη στις πιέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Κοινότητας, έχει αναθεωρήσει πλέον την νομοθεσία για την παιδική εργασία και έχει αποδεχτεί τα διεθνή πρότυπα για να οριστεί ως ελάχιστη ηλικία εργασία τα 14 έτη. Η Μογγολία έκανε μια σχετική έρευνα μετά από τη συζήτηση της σχετικής αποστολής στο πλαίσιο των γενικευμένων προτιμήσεων. Τα θεμελιώδη δικαιώματα επίσης του Κυργιστάν. Η τελευταία χώρα που μπήκε στο GSP Plus σημείωσε πρόοδο νομοθετικά σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενημέρωσε και το κατάλογο των επικίνδυνων επαγγελμάτων, προκειμένου να καταργήσει την επικίνδυνη επιθετική εργασία. Το Πακιστάν έχει εγκρίνει νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των γυναικών, σε ό,τι αφορά και τα και τις δολοφονίες τιμής. Όταν υπάρχουν επενδύσεις στις χώρες αυτές, ε, οι επιχειρήσεις μας φέρνουν μαζί τους και τα διεθνή πρότυπα, τα οποία θα πρέπει να τηρεί η εκάστοτε χώρα. Ένα άλλο στοιχείο. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται και ο επόμενος κύκλος παρακολούθησης που ξεκινάει τώρα, το 2020. Σε αυτόν τον νέο κύκλο ε, παρακολούθησης, λοιπόν, θα κοιτάξουμε κάποιους τομείς που μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Αυτά αναφέρονται και στην έκθεση. Για παράδειγμα, η ελευθερία της κοινωνίας ε, σε ό,τι αφορά την ε, λειτουργία της κοινωνίας ε, και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης μειώνονται στο Πακιστάν επίσης και σε άλλες χώρες. Επίσης γίνονται πάλι συζητήσεις για τη φανατική ποινή. Σρι Λάγκα, Μογγολία, Φιλιππίνες. Και όλο και πιο πολλές χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Γι' αυτό λοιπόν οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι σημαντικές ακόμα. Πώς λοιπόν σκοπεύουμε να εργαστούμε περαιτέρω. Εντοπίσαμε ζητήματα προτεραιότητα. Και αναχώρα επικεντρωνόμαστε σε αυτά τα ζητήματα προτεραιότητας. Αυτά θα τα βρείτε στην έκθεση ε, για την κάθε χώρα. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις αποστολές, ε, τον πολιτικό διάλογο, και να, να στέλνουμε κάθε χρόνο τα σχετικά ερωτηματολόγια. Παράλληλα, όπως είπατε, ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε και επί του μελλοντικού κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Ό,τι εμπειρίες είχαμε, τις βάζουμε στον επόμενο κανονισμό. Ό,τι μαθήματα μάθαμε. Τώρα, πριν δώσω το λόγο στην πρίση εξωτερική δράση, να πω ότι είναι, για πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά που κάνουμε αξιολόγηση και του Μπαγκλαντέ, Καμπότζη και Μιανμάρ. Ε, τις χώρες του Anything But Arms, ε, όλα εκτός από όπλα. Για την Καμπότζη θα γίνει ειδική συζήτηση σήμερα το απόγευμα. Άρα θα δούμε τα αποτελέσματα πολύ πιο λεπτομερώς. Μόλις ολοκληρώθηκε άλλωστε η αξιολόγησή μας. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλο και πιο πολύ προτίθεται να χρησιμοποιήσει το σύστημα GSP όχι μόνο να δώσει κίνητρα στις χώρες αυτές, αλλά και για να έχει δυνατότητα επιβολής κυρώσεων όταν πρόκειται για παραβιάσεις οι οποίες είναι μακροπρόθεσμες. Ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για την ενεργικό συμμετοχή του σε ό,τι αφορά το σύστημα γενικών βένων προτιμήσεων. Είναι μεγάλος ο παράγοντας μόχλαυσης που έχει το Κοινοβούλιο μέσω των επισκέψεων στις χώρες αυτές, προκειμένου να περνάμε το ίδιο μήνυμα με το μήνυμα που περνάμε και εμεί κατά τη διάρκεια τη παρακολούθηση τη διαδικασία. Ευχαριστώ και προσβλέπουμε και στη μελλοντική συνεργασία μαζί σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την υπηρεσία εξωτερική δράση, ο Γκου Χούτιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη και τη γραμματεία της ΙΝΤΑ που οργάνωσε τη σημερινή συζήτηση. Η κοινή έκθεση του 2020 που συνέταξε η Κομισιόν και ο κ. Μπορέλ, ο υπαρξεκπρόσωπος, δείχνουν την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, Απασχόληση, ε, Εργασιακών Δικαιωμάτων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και επίση ε, την εξαιρετική μόχλευση που προσφέρει αυτή η συνεργασία. Ο ύπατο εκπρόσωπος ανέφερε στι 10 Φεβρουαρίου ότι το εμπόριο είναι ένα από τα κρίσιμα εργαλεία που διαθέτει η Ένωση για να στηρίξει και να βελτιώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα εργασίας και την ε, χρηστή διακυβέρνηση που αποτελούν εργαλεία ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία έξι χρόνια το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ε, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για μας. Όταν αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ε, εργασιακά δικαιώματα είναι σημαντικά. Το GSP Plus συν το όλα εκτός από όπλα και η ενισχυμένη ε, εμπλοκή είναι σημαντικά θέματα και στοιχεία για τον πολιτικό διάλογο και τον διάλογο ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλου, για όλους όσοι παλεύουν για τα δικαιώματα και το περιβάλλον. Αυτά τα οποία λέμε στην Επιτροπή, είπαμε στην Επιτροπή όταν παρουσιάσαμε την ε, ε, έκθεση του 2018 ο ομιλητής που είναι τώρα Γενικός Διευθυντής στην απασχόληση είπε ότι τα δικαιώματα στην αγορά συνεπάγονται ε, ευθύνε και η, η τήρηση των διεθνών συμβάσεων για ανθρώπινα δικαιώματα και την εργασία είναι προϋπόθεση για να παραμείνει κανείς στο πρόγραμμα. Αυτά είπαμε το 2018 και προσυπογράψαμε μια συνθήκη, ότι η προσυπογραφή μια συνθήκης δεν σημαίνει ότι το εννοούμε. Το γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς με τι αποστολέ που στέλνετε στις διάφορες χώρες. Επιπλέον, η προόδος, νομίζω όλοι, η, πρόοδο πρόοδος κυρίως αφορά την, στα, τις διαδικασίες, δηλαδή μια βραδιπορία η GSP, το GSP sin και επίσης το EBA και το όλα εκτός από όπλα αφορούν τη μακροπρόθεσμη στήριξη αυτών που πιέζουν για την πρόοδο. Η έκθεση, όπως επίσης και το δέκατο ο έγγραφο εργασίας του προσωπικού που καλύπτει 12 χώρες δικαιούχους του GSP SYN και του όλα ε, ε, εκτός από όπλα, ε, από είναι άμεσο, ξεκάθαρο και πολλές φορές ε, αισιόδοξο, άλλες φορές όμως ε, προκαλεί στον αναγνώση αισθήματα αντιπαράθεσης και γνωρίζουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις σε πολλές από τις 71 ε, ε, υφιστάμενες χώρες. Θέματα για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, δικαιώματα μειονοτήτων, ε, θανατική ποινή και ελευθερία του συνέρχεσθε. Και ανεπαρκής πρόοδος συμπεριλαμβανομένων σε μερικές από τις μεγαλύτερες χώρες έχει αυξήσει την ε, εμπλοκή μας, κυρίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα. Όπως είπε η DG Trade της Επιτροπής, για πρώτη φορά έχουμε ένα χωριστό έγγραφο εργασίας προσωπικού για το Μπαγκλαντές, την Καμπότζη την, ε, και τη Μιαμάρ. Γνωρίζετε γιατί ξεκίνησε αυτή η ενισχυμένη συνεργασία. Αφορά τη σοβαρότητα των παραβιάσεων των αρχών ε, των συμβάσεων του ΟΗΕ και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και δεύτερον, λόγω των μεγάλων ανησυχιών σχετικά με τις παραβιάσεις αυτές που εξέφρασε ο ΟΗΕ, το ILO, η διεθνής κοινότητα συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος κοινοβουλίου και η κοινωνία των πολιτών, οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα συνδικάτα. Εν κατακλείδη, σχετικά με την έκθεση του 2020, μπορεί κανείς να πει ότι χωρίς καμία εξαίρεση οι κυβερνήσεις έδειξαν ουσιαστική συνεργασία ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σημειωθεί πρόοδος, όπως είπα πριν, βραδία, κυρίως βραδία και σε μικρές ε, σε μικρές δόσεις. Όμως ήταν χειροπιαστή και έχουμε δει βελτιώσει κυρίως όσον αφορά την παιδική εργασία. Αλλά, αλλά, πάντα υπάρχει το αλλά. Επίσης, χωρίς καμία εξαίρεση, οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά της, ε, την υλοποίηση των ε, βασικών θεμάτων. Και η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και Εργασίας έθεσαν τις προκλήσεις αυτές και τα θέματα χωρί χωρίς να χρησιμοποιούμε την βαθμολογία, τον όρο βαθμολόγηση. Αυτά τα θέματα τα θέσαμε πιο ξεκάθαρα και πιο εμφανώς στο προσκήνιο, έτσι ώστε να δοθεί μια αυξημένη ε, αίσθηση επίγοντος που θα πρέπει να καθοδηγήσει τις πολιτικές και τις δράσεις των χωρών. Πρόκειται για μια δημόσια δήλωση στην ουσία για τα όσα εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένουμε από τις χώρες αυτές ε, σε σχέση με τις μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις. Ευχαριστώ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 Um, That's not always the case when you look to a lot of the of the African countries who are lagging behind. Uh, um, uh, um, And in that sense, um, it's important that we have a very um, uh, ambitious Africa strategy. Είναι σημαντικό να έχουμε μια φιλόδοξη αφρικανική στρατηγική με αυτό το σημαντικό εμπορικό εταίρο. Θα, Δεν θα πρέπει να το λησμονήσουμε αυτό. Το θέμα της βιωσιμότητας. Η έκθεση λέει ότι μετασχηματίζονται κοινωνίες ε, ε, και μεταλαμπαδεύονται οι ευρωπαϊκές αξίες, δημιουργούνται αλυσίδε αξιών, αλυσίδες αξιών είναι σημαντικό αυτό γιατί θα πρέπει να υπάρχει κανονισμός υποχρεωτικός για τη δέουσα επιμέλεια. Ε, κάτι που ανέφερε και ο κύριος Κέλλη και οι πρόσωποι τη Κομισιόν, υπάρχουν τόσες πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρε αυτέ τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτό το πεδίο. Η Κομισιόν την περασμένη εβδομάδα ε, αφαίρεσε κάποιες, προτιμησιακές, ε, κάποιες εμπορικές ε, προτιμήσεις από την Καμπότση. Είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό της περασμένης εβδομάδας. Δεν αρκεί όμως. Θα θέλαμε να μας πει η Κομισιόν αν σκοπεύει να πάει παραπέρα. Να σας μιλήσω για δύο περιπτώσεις. Φιλιππίνες. Υπάρχουν διάφορα ανησυχητικά θέματα για τις Φιλιππίνες. Ε, πόλεμος ναρκωτικών, ε, επιθέσεις, εκτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων τον Ιούνιο τα Ηνωμένα Έθνη είπαν ότι υπήρχαν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κυβέρνηση δεν έδειξε ότι σκοπεύουν να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους για να κάνουν έρευνες σε αυτές τις περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, η αποστολή παρακολούθησης έγινε τέλη του 18 και μπορεί να μας πει η Κομισιόν να τι σκοπεύει να κάνει για να σταματήσουν οι παραβιάσει ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων στι Φιλιππίνε, Μιανμάρ. Γνωστή υπόθεση. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Δίνουμε μονομερεί ε, προτιμήσει σε χώρα που έχει κατηγορηθεί για γενοκτονία. Σοβαρέ παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρονται και συνεχίζονται. Η Κομισιόν θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν επιπλέον στοχευμένα ε, μέτρα 3,5 χρόνια μετά την αρχή της κρίσης. Ε, κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσει. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Σρι Λάνκα, γενικά, η Κομισιόν θα ήθελα να μου πει δύο πράγματα, τη γνώμη της. Πώς θα χρησιμοποιήσει τον πίνακα αποτελεσμάτων. Ε, οι εταίροι του GSP+, πώς θα δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες πληροφορίες για την εφαρμογή της σύμβασης ή των συμβάσεων και πώς θα υπάρξει ισοτιμία ανάμεσα στις μικρές δικές μας επιχειρήσεις και στις ε, ξένες ε, εταιρείες των χωρών αυτών. Περιμένουμε βεβαίω το μελλοντικό κανονισμό GSP για να δούμε περισσότερα στοιχεία. Ευχαριστώ. Από το Ρινιού, ο σκιώδη εισηγητή. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπενθυμίσατε το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων που είναι σημαντικό, προωθεί τις αξίες μας και την ανάπτυξη. Είπαν οι συνάδελφοι ότι η έκθεσή σας μιλάει για τα θετικά αλλά μιλάει και για τα προβληματικά σημεία και θα επανέλθουμε σήμερα το απόγευμα κυρίως σε μία από αυτές τις χώρες που είναι προβληματική. Επίσης, βλέπουμε την ανάγκη να παρακολουθούμε τις σχέσεις μας. Διερωτώμε λοιπόν τι ρόλο θα πρέπει να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς μπορούμε να εμπλακούμε περισσότερο ως Κοινοβούλιο. Για την έκθεσή σας, που είναι μια έκθεση που αφορά τη διετία και εγώ επειδή είμαι νέα βουλευτή, ε, επειδή έχουμε πάρα πολλέ αιτήσει εκθέσει, ε, διαρωτώ με, μήπω θα μπορούσαμε και εδώ να έχουμε αιτήσια έκθεση, γιατί έχουμε πρόβλημα να φτιάξουμε αιτήσια έκθεση και για αυτό το θέμα. Και για τη μελλοντική αναθεώρηση του συστήματο γενικευμένων προτιμήσεων. Πώς μπορούμε να εμπλέξουμε περισσότερο τις αντιπροσωπείες μας στις χώρες αυτές, γιατί αυτές μεταλαμπαδεύουν και τις ε, φιλοδοξίες μας για, ε, για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας για να πάμε ακόμα πιο μακριά για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρος, για τους πράσινους τώρα. Η κυρία Κατίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έκθεση και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά τη διάβασα με μεγάλη προσοχή. Νομίζω ότι το σύστημα από μόνο του, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων είναι πολύ επιτυχία και επιτυχές και αποτυπώνει τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς θα πρέπει να περάσει και η επόμενη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας και αυτή θα ήταν μια καλή ευκαιρία να σκεφτούμε τι μπορεί να βελτιωθεί. Δύο-τρεις ερωτήσεις έχω. Έχετε στατιστικά στοιχεία για το ποσοστό εισαγωγών ε, από τις χώρες αυτές που προέρχονται από ζώνες επεξεργασίας εξαγωγών, γιατί ξέρουμε ότι το σύστημα GSP θέλει να βελτιωθούν και οι κοινωνικές συνθήκες και οι περιβαλλοντικές συνθήκες, γιατί στις χώρες αυτές υπάρχει dumping σε ό,τι αφορά τις συνθήκες αυτές. Έχετε στοιχεία. Και τι θέλετε να κάνετε και στο μέλλον. Τα προϊόντα που έρχονται από αυτέ τι ζώνε αυτέ μπορούν μήπω να έχουν διαφορετική επισήμανση και να μην γίνονται αποδεκτά. Κατά δεύτερον, έχετε πρόβλημα, είπατε, διαφοροποίηση. Οι βασικοί τομεί είναι ο τομέα τη φαντουργία και κάποια άλλη τομεί. Πώ θα μπορούσε να μεταρρυθμιστεί το τρέχον σύστημα προκειμένου να υπάρξει οικονομική διαφοροποίηση και αυτό που είπε και ο συνάδελφο αυτό το παλιό καινούργιο φαινόμενο τη ερεκνούμενης κοινωνία των πολιτών, το οποίο επιδεινώνεται. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εφίσταμενα εργαλεία και να βελτιώσουμε τα εργαλεία που έχουμε ήδη στη διάθεσή μα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του συρρυκνούμενου αυτού χώρου. Να σα υπενθυμίσω και το ψήφισμα του προηγούμενου κοινοβουλίου, το οποίο επίσης ε, ήταν για τη μεταρρύθμιση του προγράμματο GSP και έδωσε έμφαση στη βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων. Ποιε είναι λοιπόν οι προπτικέ για τη συμπερίληψη του κλίματο και του περιβάλλοντο στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Φυσικά έχω θετική εκτίμηση για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, μονομερών προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την έκθεση ε, που είναι πλήρης έκθεση, ε, που είναι, μιλάει για κάθε χώρα. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες πτυχές της έκθεσης ε, που με προβληματίζουν και νομίζω ότι θα πρέπει να τη βελτιώσουμε δεδομένου ότι θα μεταρρυθμίσουμε και το σύστημα, να βελτιώσουμε και την έκθεση. Το 37,5% των εισαγωγών τώρα γίνονται το, με, βάση το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων plus. Είναι χαμηλό αυτό το ποσοστό, νομίζω. Βέβαια έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές, αλλά αν δείτε ε, πώς χρησιμοποιούν ε, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ε, οι χώρες αυτές, το χρησιμοποιούν μόνο ε, για δασμολογικές ποσοστώσεις. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι χαμηλό αυτό το ποσοστό. Επίσης, με τις 70, ε, ε από τις 71 ε, χώρες υπάρχουν 38 αφρικανικές δικαιούχους χώρες. Αλλά οι εισαγωγές τους είναι πολύ χαμηλές. Και εκείνοι αφορούν κυρίως τα υφοντουργικά. Επομένως, συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Κοβατσόνη. Τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να βοηθήσουμε την οικονομική διαφοροποίηση αυτών των χωρών. Δηλαδή, να αναπτύξουν και άλλους τομείς. Σε ποιο βαθμό λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα παραγωγικό ιστό και έναν επιχειρηματικό ιστό πιο ανθεκτικό και μεγαλύτερο σε αυτές τις χώρες. Για την Καμπότζη τώρα που αποφασίστηκε να αποσύρουμε τις ε, δασμολογικές ποσοστώσεις, νομίζω από το Σεπτέμβριο και μετά. Γιατί όχι πριν το Σεπτέμβριο, γιατί χρειαζόμαστε τόσο χρόνο για να μπουν σε ισχύ τα μέτρα αυτά. Η κυρία Βαν Μπρέντ μίλησε για την κατάσταση στις, Φιλιππίνες, στις Φιλιππίνες και στη Μιαμάρ. Χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα και παρόλα αυτά εποφελούνται ακόμα από το σύστημα αυτό, γενικευμένων προτιμήσεων. Δεν το αξίζουν όμως. Επίσης, οι παραβιάση ανθρωπίνων, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πότε τις εκτιμάτε υπερβολικές για να αποσύρετε το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Πρέπει να φτάσει δηλαδή η Μιανμάρ να κατηγορηθεί για γενοκτονία για να θεωρηθούν υπερβολικές οι παραβιάσεις. Επίσης, για τη μεταρρύθμιση του νέου συστήματο. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Θα ήθελα να μου πείτε το εξή. Πώ θα λάβετε υπόψη σα τι χώρε που εξακολουθούν να έχουν θανατική ποινή στην νομοθεσία τους. Δεν είναι αυτό παραβίαση ουσιαστική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ότι κάποιος δηλαδή αποφασίζει ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Για τις χώρες τώρα, οι οποίες επιβάλλουν βασανιστήρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος στην, ε, στην νομοθεσία ε, εμπόριο με χώρες χωρίς βασανιστήρια. Υπάρχει και μια πολυμερής ε, ε, πρωτοβουλία να επεκταθεί αυτό το μέτρο. Θα δώσουμε λοιπόν ε, προτιμήσεις ε, σε χώρες για να τις βοηθήσουμε να μπουν σε αυτό το σύνδεσμο χωρών που δεν έχουν βασανιστήρια. Υπάρχουν όμως χώρες μεταξύ αυτών που παρόλα αυτά έχουν βασανιστήρια και αποφελούνται από το σύστημα. Ε, ποιε είναι οι προτεραιότητέ μα, ποια είναι τα κριτήρια για να δίνουμε το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων λοιπόν σε διάφορε χώρε. Ευχαριστώ κυρία Μπρικόν. Ευχαριστώ, καλημέρα σας. Λυπάμαι που έφτασα αργά, καθυστερημένη, έρχομαι πάλι στην συνεδρίαση. Ερωτήσεις. Πρώτον, πώς μπορεί να αξιολογηθεί η θετική επίπτωση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων στο, ε, στην οικονομία της χώρας, γιατί οι εξαγωγές μιας χώρας δεν λαμβάνουν υπόψη τους ούτε την καλή υγεία της εσωτερικής οικονομίας, ούτε την κατάσταση του πληθυσμού. Ίσως με τη μεταρρύθμιση να δοθεί έμφαση στους στόχους της χιλιετίας στους στόχους της ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, η απόσυρση από την, της Καμπότζης από ένα, σύστη, από ένα μέρος του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων, μετά από αυτό το ζήτημα, το οποίο θα συζητηθεί, νομίζω ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σρι Λάγκα. Άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση της χώρας θεωρούν ότι η κατάσταση δεν έχει εξελιχθεί και δεν θα εξελιχθεί μέχρι τις ερχόμενες ε, εκλογέ. Οπότε το ερώτημα που τίθεται είναι τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι στην Σρι Λάγκα. Μήπως να χρησιμοποιήσουμε τον μπαστούνι, τις απειλές, ε, έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση των δικαιωμάτων και να σταματήσουν οι διώξεις. Ε, Τέλος, σε σχέση με αυτό που είπε και η συνάδελφος Καβατσινή ε, για τα θέματα των κοινωνικών δικαιωμάτων σε σχέση με την οικονομική κατάσταση, δεν θα θεωρούσε η Κομισιόν ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα υποβολής ε, ε, προσφυγών για τα θύματα και να υπάρχει, ας πούμε, να αυτά να λαμβάνονται υπόψη με κάποιο τρόπο. Άλλη ερώτηση. Το θέμα του φίλου συλλογικά έχουμε, ε, έχουμε δεσμευτεί να λαμβάνουμε το θέμα αυτό υπόψη μας στις εμπορικές συμφωνίες. Το θέμα το, της, βιομηχανίας ρούχων και ε, υποδημάτων που έχουν δικαιώματα εξαγωγών είναι γυναική κλάδος αυτός. Το θέμα της ε, συμπεριφοράς ε, στον, απέναντι στις γυναίκες στις χώρες εταίρους. Τέλος, το θέμα των δικαιωμάτων του παιδιού. Ίσως ε, ταχύτατα καταλήξατε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ε, πρόοδος. Βλέπουμε όμως ότι είναι μόνο έξι χώρες από τις 71. Τέλος, ε, σε σχέση με αυτό που υπόθηκε για τη Μιανμάρ. Πολλά έχουν υποθεί, πολλές εκθέσεις εδώ και χρόνια διαπιστώνουν ότι <laughs> υπάρχουν όρια και πρέπει να επιβληθούν άλλες κυρώσεις πιο περιοριστικές. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερο από αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ τρία ερωτήματα προς την Κομισιόν. Πώς ενημερώνεστε για την κατάσταση στο πεδίο. Παρήμπτος χάρη, στο Πακιστάν. Έχουμε μια εναλλακτική έκθεση ε, για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων που έχει συνταχθεί από τα συνδικάτα. Έχετε εμπλακεί στην κοινωνία των πολιτών για να καταλάβετε ουσιαστικά τι γίνεται όσον αφορά την τήρηση των, δεσμεύσεων από πλευράς χωρών. Δεύτερον, προς την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Υπάρχει τυποποιημένη μορφή ε, αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χορηγεί μέτρα ε, οικοδόμησης ε, Υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία ή εξαρτώνται τα μέτρα αυτά για την δημιουργία υποδομών από την τοπική ε, επιτροπή, ε, αντιπροσωπεία. Η, τώρα, οι χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, μερικές έχουν ε, καθεστώς χώρας όλα εκτός από όπλα και άλλες όχι. Βεβαίως αυτή είναι μια σημαντική επιτυχία, σημαντική για τις χώρες, αλλά υπάρχουν τριβές μερικές φορές μεταξύ χωρών που έχουν το καθεστώς όλα εκτός από όπλα και τους γείτονες που δεν έχουν αυτό το καθεστώς είχα μια μακρά συζήτηση με κάποιους εμπειρογνώμονες, όπως τον Πασκάλ Λαμή και άλλους. Και τελικά συμφωνήσαμε να ζητήσουμε να χορηγηθεί το καθεστώς όλα εκτός από όπλα σε όλες τις χώρες στην υποσαχάρη Αφρική. Τι γνώμη έχετε από αυτού. Okay, let me cover some of the... Θα καλύψω μερικά από τα ερωτήματα, θα τα συγκεντρώσω. Κάποιες από τις ερωτήσεις ήταν ε, ταυτόσιμες ε, από διαφορετικούς δηλαδή βουλευτές. Είχαμε τις χίλιες ερωτήσεις, οπότε θα τις αμοδοποιήσω τις απαντήσεις. Για το σύστημα. Και πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε ορισμένε χώρες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Είναι προβλήματα που έχει εντοπίσει η διεθνή κοινότητα και οι διεθνεί φορεί παρατήρησης. Αναφέρθηκε η Μιανμάρ, η Σρι και οι Φιλιππίνες. Ξέρουμε πολύ καλά την κατάσταση και στις τρεις χώρες. Και μεταχειριζόμαστε και αντιμετωπίζουμε την κάθε χώρα διαφορετικά, ανάλογα με τα δεδομένα της. Η Μιανμάρ ε, επιλέγει για να έρθουμε σε επαφή Έχουμε επιταχύνει και πολλαπλασιάσει τις συζητήσεις με την κυβέρνηση, έχουμε κάνει επισκέψεις, εκτεταμένες συζητήσεις, έχουμε στείλει ερωτηματολόγια ε, και δελτία και πιέζουμε ήπια για να υπάρξει αλλαγή. Θέλουμε μια μεγαλύτερη αλλαγή. Θα θέλαμε μάλλον, αλλά είναι δύσκολο, γιατί είναι θέμα κουλτούρας, ε, θέμα μειονοτήτων και πώς τις βλέπουν. Ε, επίσης, ε, το πολιτικό καθεστώς που ξέρετε ότι τις αποφάσεις τις παίρνει ο στρατός. Το φθινόπωρο θα γίνουν εκλογές στη Μιανμάρ, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη συνολική κατάσταση και δεν θέλουμε να επιτείνουμε τις συγκρούσεις. Θέλουμε να τις ελαφρύνουμε και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο όπου μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος. Επομένως, σχεδιάζουμε να κάνουμε μια άλλη επίσκεψη πριν τις εκλογές για να προσπαθήσουμε να πιέσουμε για κάποια θέματα. Ε, και δεν είναι μόνο η είναι και άλλα θέματα που μας απασχολούν. Είναι η εκπαίδευση. Ε, ε, είναι τα θέματα των εσωτερικά εκτοπιστέντων. Είναι μακρύς ο κατάλογος, αλλά η πρόκληση είναι τεράστια. Δεν είναι μόνο το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Επίσης, υπάρχουν ε, ευθύνες και στα κρατη Να είναι πολύ πιο φιλόδοξα για το πώς θα αντιμετωπίζουν τη χώρα αυτή, τη Μιανμάρ. Φιλιππίνες και Σριλάνκα τώρα. Και αυτές οι χώρες είναι στον κατάλογό μας. Πρέπει να τις ελέγξουμε πολύ περισσότερο έχουμε μία βαθμία προσέγγιση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μία ισορροπία ανάμεσα στη διατήρηση του διαλόγου, να κρατήσουμε την πόρτα ανοιχτή για συζήτηση, να συνεχίσουμε όμως την πίεση και να μην καταστρέψουμε όλες τις γέφυρες που έχουμε χτίσει με αυτές τις χώρες. Συχνά στις επισκέψεις μας διαπιστώνουμε ότι έχουμε προοδευτικές δυνάμεις στη χώρα και μπορούμε να ενισχύσουμε αυτές τις προοδευτικές δυνάμεις. Ε, αναφερθήκατε σε παράλληλη, ε, παράλληλες εκθέσεις ε, στο Πακιστάν που χρηματοδοτούμε εμείς. Στο ε, μπορεί δεν έχουμε δυνατότητα χρηματοδότησης, αλλά στηρίζουμε αυτές τις, τα συνδικάτα και τις ΜΚΟ για να διαδώσουμε τις πληροφορίες για το πώ λειτουργεί το σύστημα γενικευμένων αποτιμήσεων, για να διορθώσουμε τι παράλληλε εκθέσει, για να τι ενισχύσουμε, για να μπορούν να συζητούν αυτέ οι οργανώσει ε, και αυτά τα σωματεία ε, με την κυβέρνηση απευθεία. Επίση, προσπαθούμε να δούμε ποιε είναι οι πηγέ πληροφορίας. Για μα είναι οι φορεί ε, παρακολούθηση του ΟΗΕ και του Διεθνού Γραφείου Εργασία. Και οι δύο οργανισμοί μας έδωσαν ανησυχητικέ εκθέσεις για καταστάσεις σε αυτές τις χώρες και τις εξετάσουμε πολύ πιο προσεκτικά. Ένα άλλο θέμα για... αφορούσε το ρόλο του Κοινοβουλίου. Το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων προϋποθέτει συλλογική προσπάθεια Κομισιόν, Κοινοβούλιο και κρατημέλη. Είμαστε έτοιμοι για να ερχόμαστε εδώ πάντα συνεδριάσει, να ενημερώνουμε του ευρωβουλευτέ αν επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για κάποια συγκεκριμένη χώρα, είτε κυκλισμένων των θυρών, είτε σε δημόσια συνεδρίαση. Πάντα είμαστε στη διάθεσή σας και πιστεύουμε ότι πρέπει να στέλνουμε τα ίδια μηνύματα όλοι μας σε αυτές τις χώρες. Ότι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες, τις ίδιες προτεραιότητες, για να το πω έτσι. Καμία από αυτές τις χώρες δεν είναι τέλεια. Όλες είναι περιπροκές χώρες σε ό,τι αφορά την πολιτική δυναμική τους και την οικονομική ανάπτυξή τους, αλλά θα πρέπει να εστιάζουμε εκεί που μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Αλλιώς, σπαταλούμε τους πόρους μας. Λοιπόν, συμπιέζονται οι ΜΚΟ, το ξέρουμε, το παρατηρήσαμε, Αφρική. Μία-δύο ερωτήσεις ακούστηκαν για την Αφρική. Τι θα γίνει με αυτή την Ήπειρο. Πρέπει να ομολογήσω ότι μέχρι στιγμής δεν είχαμε εστιάσει πολύ στην Αφρική. Δεν είχαμε τους πόρους, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Ασχολήθηκαμε με το GSP+, γιατί είναι χώρες που όταν μπήκαν σε αυτό το σύστημα, ε, είχαν αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις για συνεργασία. Ε, μας επέτρεψαν να πάμε στη χώρα τους. Ε, ετοίμασαν εκθέσεις προς εμάς. Ε, για το Everything But Arms ε, διαλέξαμε το Bangladesh, Μιανμάρ και Καμπότζη για αυτές τις χώρες, ε, σε αυτές τις χώρες ε, εστιαστήκαμε, γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, αλλά και λόγω του επίπεδου εμπορίου που έχουμε. Ε, ερώτηση για το 36%. Πώς ε, δικαιολογούμε το εμπόριο. Και γιατί το λέμε επιτυχές μια και μόνο το 36% του συνολικού εμπορίου συνδέεται με το GSP. Το να, το να οι εισαγωγέ ε, χωρί δασμού είναι πολύ περισσότερα προϊόντα. Μερικέ φορέ είναι 100%. Απλώ δεν αναφέρεται ω GSP. Ε, οι περισσότερες αφρικανικές χώρες εξάγουν ε, ορυκτά και πρωτεσίλες που έρχονται με μηδενικούς δασμούς στην Ευρώπη ούτως ή άλλως. Είναι ε, οι δασμοί του πλέον ευνοούμενου κράτους. Συνολικά, οι περισσότερες λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ε, κατά 80-90% εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αδασμολόγητα, δηλαδή χωρίς, μπαίνουν τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ, χωρίς καθόλου δασμού. Ένα άλλο ερώτημα. Επομένω, η Αφρική, ναι, δεν την ξεχνάμε, την έχουμε στο μυαλό μας για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις επαφές. Υπάρχει όμως και μια άλλη προσπάθεια που γίνεται, η Συμφωνία οικονομική εταιρική σχέση. Έχουμε και διμερείς επαφές όπου προσπαθούμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις μας για ζώνες ελευθέρου εμπορίου. Για συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Για την ΕΠΑ και την αν μπορούμε να επεκτείνουμε το Everything But Arms ε, και σε άλλες χώρες. Ε, έχουμε ένα καθεστώς που βασίζεται σε κανόνες. Μία χώρα παίρνει το όλα πλην όπλων εφόσον είναι λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα. Εάν δεν είναι λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα, και υπάρχουν μερικέ χώρε στην Αφρική που δεν είναι, δεν μπορούμε να του δώσουμε αυτό το καθεστώ ε, όλα πλην όπλων. Δεν το ξέρω. Ναι, μετά... Φυσικά θα συζητήσουμε κατά πόσο είναι δυνατόν ή δεν είναι δυνατόν να δοθεί αυτό το καθεστώ ε, σε όλες τις υποσαχάριες χώρε. Είμαι πεπισμένο ότι νομικό αυτό είναι δυνατόν. Θα γίνει συζήτηση για το GSP και για το θέμα της Αφρικής. Από πλευρά τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι δικαίωμα του Πρόεδρου να απαντήσουμε πρώτα στη δική σα ερώτηση σε ό,τι αφορά την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Εγώ ο ίδιος ε, πρέπει να πιστοποιήσω γιατί έχω μεταβεί σε πολλές αποστολές ε, και στην Καμπότζια, στο σύστημα όλα εκτός από όπλα και στο GSP+. Πριν, ε, κατά τη διάρκεια και μετά τις αποστολές, συμμετείχαμε σε συζητήσεις με την κοινωνία των πολιτών και εκπροσώπους εδώ στις Βρυξέλλες για να κανονίσουμε μετά το ταξιδιού και επιτόπου με τις απαραίτητες προφυλάξεις σε ό,τι αφορά την ε, εμπιστευτικότητα. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής έθεσε το ερώτημα για την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία. Η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία συμμετέχει σε κάποιες περιπτώσεις ως πρώτη αρχή κατάρτισης των εκθέσεων, των ε, ε, τήσιων εκθέσεων και βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό στις πηγές ε, του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας και της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας εκεί. Σε ό,τι αφορά την τρίτη έκθεση τώρα, διαπιστώνουμε μεγαλύτερη προσοχή από όλα τα μέλη και τους επικεφαλείς αντιπροσωπιών στις χώρες GSP Plus και όλα εκτός από όπλα. Δεν είμαστε ακόμα σε τέλειο επίπεδο, αλλά πάμε καλά. Ε, για την ανάπτυξη τώρα υποδομών, το capacity building, να πω ότι υπάρχει στενή σύνδεση όλων των προγραμμάτων για την ανάπτυξη δυναμικού σε ό,τι αφορά και τους στόχους για την ε, ανάπτυξη, τα ευρωπαϊκά, τα δικαιώματα των πολιτών τα κοινωνικά δικαιώματα και σε ό,τι αφορά και την Υποεπιτροπή Καλή Διακυβέρνηση για κάποια άλλα ερωτήματα τώρα που ακούσαμε. Νομίζω ότι το είπαμε και προηγουμένω ε, ω υπηρεσία εξωτερική δράση ότι είναι καλό το GSP. Αλλά δεν είναι και σουητικό σουγιάς όπως είπε και η Επιτροπή, δεν επιλύει αυτό όλα τα προβλήματα σε όλες τις χώρες. Πολλά εξαρτώνται από τις άλλες πολιτικές, από την εξωτερική πολιτική, τα μέτρα περιοριστικά, την ανάπτυξη δυναμικού. Και προφανώς η έκθεση δεν έχει να κάνει με την ταξινόμηση των χώρων που ωφελούνται από το GSP Plus και το εκτός από όπλα ή να συστήσουμε περαιτέρω προνομιακή μεταχείριση. Αλλά φυσικά έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα, αν τα πράγματα χειροτερεύσουν και επιδεινωθούν σημαντικά, να αφαιρέσουμε κάποια προνόμια. Να αναφέρω και αυτό που είχε πει ο Μπορέλ όταν έλευθε η απόφαση για να αφαιρεθούν τα προνομία από την Καμπότζη. Είχε πει τότε ότι η διάρκεια, η κλίμακα και ο αντίκτυπος της παραβίασης του δικαιώματος πολιτικής συμμετοχής και της ελευθερίας συντηρίζεσθε και ε, ελεύθερης έκφρασης ε, στην Καμπότζη δεν άφηνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλα περιθώρια παρά να αποσύρει το καθεστώς αυτό. Όταν διαβρώνονται λοιπόν τα δικαιώματα και η δημοκρατία, όταν καταπνίγεται ο ελεύθερος διάλογος, αυτά συμβαίνουν. Δεν υπάρχει απόλυτος αυστηρός κανόνα ε, σε, σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το τι αποτελεί και συνεπάγεται μια συστηματική και κατάφορη παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά το GSP Plus και τους ε, χώρες που οφειλούνται. Υπάρχει ένα περιθώριο ευχέρειας. Από πλευρά του Κοινοβουλίου έχω να πω ότι αποτελείται ένα από τα βασικά θεσμικά όργανα που θα μας καθοδηγήσετε σχετικά με το πότε έχει υπερβληθεί ένα όριο. Μία ερώτηση που έγινε για τις Φιλιππίνες. Είπα και προηγουμένως ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι εκθέσεις πραγματικά είναι συνταρακτικές. Κοιτώντας τη σελίδα 1 της έκθεσης, δεν ε, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, αυτό που αναφέρεται για την θανατική ποινή για τέτοια εγκλήματα. Αν αυτό επανεισαχθεί, θα αποτελέσει παραβίαση του δεύτερου συμπληρωματικού εθελούσιου πρωτοκόλου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι κάτι πολύ ξεκάθαρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα, έχει δώσει σαφείς ε, ενδείξεις για το τι θα συμβεί αν περάσει αυτό. Θα ήταν ε, αντίθετο με το πνεύμα της ε, Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού. Επίσης, ακούσαμε και ερωτήματα για τη Μιαμάρ. Αν ένα πράγμα μπορούμε να πούμε για την κυβέρνηση αυτή, είναι το εξή. Είναι ότι έχει δεσμευτεί. Σοβαρά. Τώρα μπορεί να ρωτηθεί κανεί ε, πιο μέρος της κυβέρνηση. το πολιτικό σκέλο. Είχαμε όμως και επαφέ και με το στρατιωτικό σκέλο της κυβέρνηση εν μέρη. Αλλά η μερική πρόοδο αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο είναι δεδομένο. Για την επικύρωση επίσης ε, της σύμβασης 138 του ΠΟΕ για την, ε, τα ιστορικά εκτοπιστέντα άτομα έχει ψηφιστεί σχετικό νόμο Πολλά άλλα προωθούμε και η ανθρωπιστική ε, πρόσβαση σε κράτη στο εσωτερικό της χώρας. Και επίσης σε ό,τι αφορά την εισαγωγή προσωρινών μέτρων και τη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τις Φιλιππίνες και πάλι. Έχουμε μια υποεπιτροπή για την καλύτερη κυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πριν από δύο εβδομάδες ε, ιδρύθηκε. Δεν έχει ακόμα γίνει συνεδρίαση, αλλά υπάρχει αυτή η υποεπιτροπή. Υπάρχει λοιπόν μία πρόοδος. Θα έλεγα έξι πλήν, τουλάχιστον αν με ρωτούσατε να κάνω μια ταξινόμηση. Δεν μιλάμε για τις χώρες οι οποίες έχουν κορυφαία δέσμευση και ανταπόκριση σε αυτά που ζητάμε. Δύο λεπτά, δώστε μου να κοιτάξω και τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Την δέωση επιμέλεια. Να υπενθυμίσω το σημείο αυτό, το εξή. Γίνονται σχετικέ ε, έρευνε, Η Γενική Διεύθυνση δικαιοσύνη, ε, κοιτάει το θέμα τη δεωση επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού. Να πω κάτι ξεκάθαρα. Η πρόσβαση σε συλλογικά ένδικα μέσα δεν αποτελεί στοιχείο δέουσας επιμέλειας. Όπως αναπτύσσεται μπορεί να προσθεθεί από τις εταιρείε, αλλά η δέουσα επιμέλεια αφορά τις εταιρικέ διαδικασίες εθελούσες ή υποχρεωτικές για να ξέρουμε πώς αντιμετωπίζουμε κάποιους κινδύνους προκειμένου να λάβουν μέτρα για την ε, επίλυση των ζητημάτων. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Μπορεί να μου έφυγαν και δύο-τρία στοιχεία. Αν κάτι παρέλειψα, παρακαλώ να μου το υπενθυμίσετε, αξιότιμοι βουλευτέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Λίκη Πρόεδρο. Ευχαριστώ, κυρία Καβατσίνη. Δεν ε, ε αναφερθήκατε στα EPZ. Δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε στατιστικά στοιχεία για αυτά. Τα, στοιχεία είναι απόρριτα και καταγεγραμμένα για όλη τη χώρα. Αλλά η γενική προσέγγιση μας είναι η εξή. Η ευθύνη διατήρησης των προτύπων στον τομέα αυτό ανήκει στη χώρα και η χώρα λογοδοτεί στους διεθνείς οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων και του EPZ. Δεν μπορούμε λοιπόν να ενθαρρύνουμε ούτε καν ε, θεωρούμε ότι είναι δυνατόν τα επίπεδα αυτά, τα πρότυπα αυτά να είναι χαμηλότερα ή να αντιβαίνουν σε αυτά τα οποία προβλέπει ο ΟΗΕ και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Ε, λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό γιατί το επόμενο θέμα είναι και κλεισμένων των θυρών, οπότε σας παρακαλώ να ε, όσοι δεν θα παραμείνουν να... Ε,